Είναι περασμένες οι τρεις, οπότε μπορούμε να ξεκινήσουμε. Ε, το πρώτο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι ε, ε, εκλογή του Προέδρου, αλλά νομίζω πως είναι για να πρόκειται για σχέδιο της ημερήσιας διάταξης, γιατί εγώ ακόμα εδώ είμαι. Τέλος πάντων, θα το θυμάμαι. Πάντως θυμάμαι, Κλάουδιο, ότι μου είχε πει ότι είπες ότι ε, το Brexit είναι σαν να βρίσκεται κανείς, σαν να είναι καταδικασμένος σε θάνατο και να περιμένει την εκτέλεσή του. Οπότε, εν πάση περιπτώσει, κάπω έτσι είναι η κατάστασή μου. Σε κάθε περίπτωση όμω χαίρομαι που θα είμαι εδώ μαζί σα για τι επόμενε εβδομάδε. Έχουμε εδώ νομίζω μια ομάδα από τη γερμανική τηλεόραση. Έτσι εδώ σε κάποια απόσταση από εμά. Ωραία. Άρα λοιπόν, το πρώτο σημείο είναι η έγκριση τη ημερήσια διάταξη. Επειδή μα ζήτησε αύριο να κάνουμε μια μικρή αλλαγή στην ημερήσια διάταξη σε ό,τι αφορά ε, την ετήσια έκθεση για τον αλληλευτικό στόλο μα και το να εξετάσουμε δηλαδή αυτό το ζήτημα πριν από τον τεχνικό πτυρωτών. Ε, νομίζω πω δεν είναι μεγάλη αλλαγή, οπότε ελπίζω να μπορείτε να συμφωνήσετε όλοι με αυτό. Εάν ε, μπορούμε να το κάνουμε έτσι, περνάμε στην έγκριση των ε, πρακτικών της, ε, των συνεδριάσεων τη 24 η Σεπτεμβρίου και της Δευτέρα και 3ης Οκτωβρίου. Εάν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, θεωρούμε πως εγκρίνονται και αυτά τα πρακτικά. Υπό το σημείο 3 η δηλαδή ανακοινώσει του Προέδρου, δεν υπαρχουν αντιρρησει θεωρουμε πω εγκρινονται και κάτι ιδιαίτερο από την πλευρά μου. Οπότε περνάμε στο πρώτο ουσιαστικό σημείο της ημέρας σας διάταξης για σήμερα που είναι η παρουσίαση μιας έκθεσης από την Διακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή μια έκθεση σε ό,τι αφορά ε, τους ωκεανούς και την κρυόσφαιρα σε ένα μεταβαλλόμενο κλίμα. Ε, θα έχετε παρακολουθήσει ε, κάποια από σας συζητήσεις που έγιναν στο επίπεδο της Επιτροπής ΕΝΒΗ σε σχέση με αυτό το ζήτημα και μα ενδιαφέρει βέβαια ιδιαίτερα εδώ το σχετικό ζήτημα από την οπτική γωνία τη Αλία. Οπότε θα ήθελα να ε, καλωσορίσω εδώ τον ε, καθηγητή, τον ε, Δ. Hans Otto Pörtner, που είναι ο συμπρόεδρος της ομάδας εργασίας 2, αν δεν με της IPCC, έτσι ώστε να μας παρουσιάσει την οπτική γωνία ακριβώς της IPCC σε σχέση με αυτό το ζήτημα. Παρακαλώ κύριε Πέρτνερ, έχετε το λόγο. Ναι, σας ευχαριστώ πολύ. Ξεκινάμε εδώ με ένα τρέλερ λοιπόν. The frozen parts of the world.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 Together, we can build a sustainable and equitable future for all. Our future is in our hands. Yeah, we set little uh, trailer. Είδαμε λοιπόν ένα μικρό ε, τρέλερ. Σας ευχαριστώ λοιπόν που μου δίνετε τη δυνατότητα σήμερα να σας κάνω μια παρουσίαση σε ό,τι αφορά τα κύρια απόρρισματα αυτή τη έκθεσης της ε, IPCC σε ό,τι αφορά τους ωκεανού ε, και την κρυόσφαιρα σε ε, ένα μεταβαλλόμενο κλίμα. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν εδώ με την παρουσίαση PowerPoint στι οθόνε. Θα σας παρουσιάσω το σύνολο της έκθεσης, αλλά θα εστιάσω ειδικότερα στο κομμάτι των ωκεανών. Ε, και όπως βλέπετε εδώ και από την αρχική διαφάνεια εξετάζουμε τα βουνά με υψηλό ισόμετρο, τις επολικές περιοχές και συνέχεια εξετάζουμε την θάλασσα, τους ωκεανούς δηλαδή γενικότερα και τις επιπτώσεις που όλα αυτά έχουν ε, με την αλλαγή του κλίματος για την ε, θαλάσσια ζωή.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 I see that struggling with technology can even happen at EU e level. Okay, Ωραία, λοιπόν λύθηκε το πρόβλημα, επιστρέφω στην έκθεση. Άρα λοιπόν ε, στον πυρήνα εδώ της έκθεσης βρίσκονται οι ωκεανοί και όπως βλέπετε στην αρχική διαφάνεια εδώ, στην αρχική σελίδα της έκθεσης εδώ έχουμε να κάνουμε με τις επιπτώσεις κλιματικής αλλαγής σε όλα τα υψόμετρα και το πώς ε, σταθεροποιεί ουσιαστικά ο ωκεανός το ε, σύνολο εδώ του θέμα του πλανήτη. Ε, αυτή η έκθεση λοιπόν αποτέλεσε το αποτέλεσμα εντατική εργασία επί σειράς τριών ετών και ήμασταν συνολικά 104 συντάκτες, των οποίων το 31% ήταν γυναίκες. Από 36 συνολικά χώρες συντάκτες και είχαμε 6.980 μελέτες επιστημονικά δηλαδή έγγραφα και ε, ακριβώς επειδή ε, προσέλκυσε τόσο μεγάλη προσοχή ε, ως επιστημονικό ε, πόνημα υπήρξαν συνολικά 31.176 ε, σχόλια. Ποιο είναι όμως το βασικό μήνυμα αυτής της έκθεσης, ότι η ωκεανοί και η κρυόσφαιρα του πλανήτη πραγματικά ε, έχουν δεχτεί ε, ισχυρέ πιέσει από την κλιματική αλλαγή ε, επί σειρά δεκαετιών και οι επιπτώσεις για τη φύση και την ανθρωπότητα είναι σαρωτικές και πολύ σοβαρές. Ξεκινάμε εδώ λοιπόν από τα βουνά σε ψηλό υψόμετρο και το λιώσιμο εδώ των παγετών, πράγμα το οποίο θα έχει απρόβλεπτες συνέπειες, ειδικότερα και για τους ανθρώπους οι οποίοι διαβιούν στι σχετικέ περιοχέ. Μιλάμε δηλαδή για 700 εκατομμύρια συνολικά ανθρώπου, οι οποίοι θα μπορούσαν δυνητικά να υποστούν τι συνέπειε από το λιώσουμε αυτών των ε, παγετών. Μετά περνάμε στις πολιτικές περιοχές, δηλαδή εξετάζουμε εδώ και την Αρκτική και την Ανταρκτική. Και ε, ποια είναι τα βασικά μηνύματα της έκθεσης σε σχέση με αυτές τις πολιτικές περιοχές, ότι η τα στρώματα πάγου στη Γρυλανδία και στην Ανταρκτική μειώνονται σε όγκο. Ε, αυτό σημαίνει αύξηση τη ε, στάθμης ε, τη θάλασσα, θα συνεχίσουν μάλιστα να λιώνουν και αυτό σημαίνει ότι θα υπάρξει και μακροπρόθεσμη άνοσμος τη στάθμης τη θάλασσα. Και επίση ε, οι πάγοι στις θάλασσες τη Ακτική μειώνονται όλο ένα και περισσότερο, χάνουν και σε πάχο και εάν έχουμε την θέρμανση του πλανήτη κατά 1,5 ε, βαθμό ο Αρκτικός ωκεανός ε, ουσιαστικά ε, κάποιες στιγμές ε, δεν θα υπάρχει καθόλου πακέτο στον Αρκτικό ωκεανό ενώ σε θέρμανση με κατά δύο ε, βαθμούς Κελσίου αυτό δηλαδή το να μην υπάρχουν επαγγελίες, μπορεί να συμβαίνει ένα χρόνο ανα, κάθε τρία χρόνια. Ταυτόχρονα η μόνιμη παγετή λιώνουν όλα και περισσότερο και αυτό που σημαίνει ότι μπορεί να αυξήσει σε περισσότερες εκπομπές αερίων του θερμοτυπίου και ε, εάν οι εκπομπές ε, συνεχίσουν να αυξάνονται γύρω στο 70% της, ε, των μόνιμων παγετών που βρίσκονται κοντά στα στάθμη της θάλασσας θα εξαφανιστούν. Και εδώ βέβαια θα υποστούν τι συνέπειε οι άνθρωποι οι οποίοι ζουν στι αρκτικέ περιοχέ, οι ταγενεί δηλαδή ιδιαίτερα, και ήδη προσαρμόσουν του τρόπου με του οποίου κυνηγούν, με του οποίου μετακινούνται στην εποχικότητα και στην ε, ασφάλεια βέβαια των παγετών και των ε, γενικά τη κατάσταση των καιρικών συνθήκων και ε, το κατά πόσο θα μπορέσουν να προσαρμοστούν επιτυχώ θα εφαρμοστεί και από τι δυνατότητε χρηματοδότηση και τι σχετικέ ικανότητε. Τώρα, περνάμε στου ωκεανού και την θαλάσσια ζωή και το ποιε είναι οι επιπτώσει τη κλιματική αλλαγή. Όπω σα είπα, ήδη οι ωκεανοί έχουν απορροφήσει περισσότερο από το 1% της ε, αυξημένης ε, θερμοκρασίας στο κλιματικό σύστημα και έως το 2100 ε, οι ωκεανοί θα έχουν απορροφήσει 2-4 φορές περισσότερη θερμότητα από την παγκόσμια θέρμανση εάν περιοριστεί η συνολική θέρμανση σε 2 βαθμούς, ενώ θα μπορούσε να είναι πολύ ψηλότερο αν έχουμε υψηλότερη αύξηση. Και επίση βέβαια αυτή η αύξηση τη θερμοκρασία των ωκεανών σημαίνει μικρότερη μίξη των στρωμάτων της ε, θάλασσας και αυτό σημαίνει λιγότερο οξυγόνο για την θαλάσσια ζωή. Επίσης, τα νήματα θερμότητα ε, στη θάλασσα γίνονται όλο και πιο ισχυρά, που σημαίνει ότι μπορεί να υπάρξουν αντικές συνέπειε ε, για τα κοράλια, για φύκια και ούτω καθεξής. Και επίσης βλέπουμε με την περισσότερες εκπομπές άνθρακα τις οποίες απορροφούν οι ωκεανοί, έχουμε περισσότερη οξύνση των ωκεανών. και αυτό βέβαια με, τις, με την παραμονή αυτών των εκπομπών θα συνεχίσει να επιδεινώνεται. Ας ε, δούμε λοιπόν ε, το τι συμβαίνει εδώ σε ό,τι αφορά δηλαδή την ε, φυσική και την χημεία στους ωκεανούς. Βλέπουμε δηλαδή τι θα μπορούσε να συμβεί σε περίπτωση όπου παραμείνουν οι εκπομπές και οι συνθήκες γενικά ότερα όσο έχουν ή φιλόδοξη μείωση των εκπομπών όπου θα φτάναμε δηλαδή σε θέρμανση κατά 1,5 βαθμό Κελσίου. Δηλαδή εκεί θα είχαμε σταθεροποίηση της κατάστασης. Στα αριστερά λοιπόν βλέπουμε την ε, θερμοκρασία σε ό,τι αφορά τον ε, αέρα δηλαδή, τους, τις μέσες θερμοκρασίες και μετά ε, την θερμοκρασία στην επιφάνεια της θάλασσας η οποία υστερεί λίγο σε σχέση με τον αέρα οι μέρε όπου θα υπάρχουν αυτά τα απονομενόμενα heat waves, ε, δηλαδή περίοδοι ιδιαίτερης, ε, ιδιαίτερα υψηλή θερμοκρασία στους ωκεανού, θα αυξάνονται όλο και περισσότερο. Αντιθέτω, εάν υπάρξουν ε, φιλόδοξοι στόχοι που θα επιτευχθούν σε ό,τι αφορά τη μείωση των εκπομπών, θα επιτευχθεί σταθεροποίηση. Ε, στα δεξιά βλέπουμε τώρα κάποιε ε, ε, χημικές παραμέτρους, δηλαδή σε ό,τι αφορά το pH στην Ε, το pH δηλαδή στους, ε, στην επιφάνεια των ωκεανών και πώς μπορεί να σταθεροποιηθεί. Επίσης, ε, μόλις σας παρουσίασα ότι υπάρχει και επίπτωση από την κλιματική αλλαγή στη διαθεσιμότητα οξυγόνου. Και ενώ έχουμε μια πιο ήπια εικόνα όταν έχουμε το σύνολο των ωκεανών. Υπάρχουν κάποιε περιοχέ οι οποίε ήδη έχουν χαμηλότερα επίπεδα οξυγόνου και εκεί θα μπορούσαμε να έχουμε πολύ ε, σοβαρέ ε, συνέπειε. Και ε, μετά βλέπουμε και πάλι τις δύο, τα δύο διαφορετικά σενάρια στο τελευταίο γράφημα κάτω δεξιά σε ό,τι αφορά δηλαδή την ε, έκταση των πάγων στην Αρκτική θάλασσα. Τώρα, έχουμε από τη μία κάποια δεδομένα τα οποία έχουμε παρατηρήσει και από την άλλη πλευρά έχουμε ε, κάποιες προγνώσεις. Δηλαδή, καταρχήν έχουμε κάποια βασικά δεδομένα που τα βλέπουμε εδώ σε κίτρινο και σε πράσινο χρώμα και μετά τα υπόλοιπα όπου εστιάζουμε σε πολύ, ε, σε πολύ συγκεκριμένα δεδομένα ε, σε ό,τι αφορά δηλαδή για παράδειγμα κοράλια, ε, φύκια, ε, βενθοπελαγικές ε, περιοχές και ούτω καθεξής. Και από εκεί και μετά το πώς επηρεάζονται άλλοι τομείς όπως για παράδειγμα της αλληλείας, του τουρισμού, των μεταφορών και ούτω καθεξής. Και για πολλές από αυτές τις παραμέτρους βλέπουμε κάποια αύξηση για παράδειγμα σε ό,τι αφορά τη θερμοκρασία ενώ μείωση για παράδειγμα του pH. Και βλέπουμε ακριβώς πώς καταδεικνύεται εδώ η επίπτωση και το πόσο τελικά είναι αρνητική οι αρνητικές οι συνέπειες της ε, θέρμανσης ε, των ωκεανών ε, για την θαλάσσια ζωή και τα σχετικά οικοσυστήματα. Και το, τα πιο ευάλωτα οικοσυστήματα τα οποία αναγνωρίσαμε σε αυτή την έκθεση σε σύγκριση και με τον τελευταίο κύκλο αξιολόγησης δηλαδή τον 1,5 γιατί είμαστε ήδη στον έκτο κύκλο είναι λοιπόν η κορελογενής ύφαλη σε θερμά ύδατα. Και βλέπουμε δηλαδή την φωτογραφία όπου ουσιαστικά υπάρχει λεύκανση αυτών των κορελογενών υφάλων ακριβώς επειδή ε, υπάρχουν αρνητικές επιπτώσει σε ό,τι αφορά την φωτοσύνθεση. Και όταν δηλαδή υπάρχει μια τέτοια ε, ε παρατεταμένη περίοδος ε, υψηλής θερμοκρασίας στον ωκεανό δεν είναι δυνατή, ε, μπορούν ε, τα κοράλια να απορροφήσουν τα άλγη τα οποία χρειάζονται για τη φωτοσύνθεσή τους και πεθαίνουν στη συνέχεια όπως βλέπουμε για παράδειγμα στην φωτογραφία στα δεξιά. Βλέπουμε τώρα εδώ στο γράφημα μια σχετική ποσοτικοποίηση αυτών των, ε, των επιπτώσεων, δηλαδή των επιπέδων κινδύνου και διαπιστώνουμε δηλαδή όπου υπάρχει κόκκινο χρώμα ότι ήδη έχουμε ξεπεράσει τα επίπεδα απόλυτου κινδύνου. Ανάμεσα δηλαδή στα χρόνια 2006-2015. Και πάντοτε εδώ βασιζόμαστε στον μέσο όρο της ε, θερμοκρασίας στην επιφάνεια ε, των ωκεανών. Και βέβαια εστιάζουμε στον στόχο του 1,5 βαθμού Κελσίου και για τον οποίο βασιστήκαμε και στην παγκόσμια έκθεση σε ό,τι αφορά ακριβώ αυτό το σενάριο τη θέρμανση κατά 1,5 βαθμό Κελσίου. Και στι τρει ειδικέ εκθέσει, δηλαδή τι οποίε ε, ήδη έχουμε πονήσει στο πλαίσιο αυτού του κύκλου εργασιών, έχουμε πάντοτε βασίσει σε αυτό το 1,5 βαθμό. Και βλέπουμε λοιπόν σε ό,τι αφορά τα κοράλια στα θερμά ύδατα έχουμε ήδη και στον 1,5 βαθμό ε, πολύ ε, αρνητικέ ε, συνέπειε. Ενώ αντιθέτω, για παράδειγμα, στα μάγκροβ, τέτοιου είδου δηλαδή υγροτόπου, έχουμε πολύ χαμηλότερε επιπτώσει, λιγότερο σοβαρέ. Και σε ό,τι αφορά τις, την αλληλεία μικρής κλίμακας, ειδικότερα σε χαμηλά υψόμετρα, έχουμε και σε χαμηλά επίπεδα, συγγνώμη, έχουμε και πάλι πολύ σοβαρέ συνέπειε με βάση το 1,5 του 2 Κελσίου. Εδώ σε ό,τι αφορά του κοραλογενούς φάλους ακόμα και αν παραμείνουμε στον 1,5 βαθμό ε, Κελσίου υπάρχει πολύ ψηλό κίνδυνος να χάσουμε 70 90% των κοραλογενών υφάλων και τα σχετικέ ε, υπηρεσίε ε, για την ανθρωπότητα. Άρα λοιπόν το συμπέρασμα είναι ότι ήδη υπάρχει σοβαρή θύρμανση και ήδη υπάρχουν πολύ σοβαρές συνέπειες με αποτέλεσμα να καταστρέφεται ένα πολύ σημαντικό κομμάτι των θαλάσσιων οικοσυστημάτων. Τώρα, κάναμε μια αξιολόγηση στο πλαίσιο αυτή τη έκθεση και για πολλά άλλα οικοσυστήματα. Βλέπουμε εδώ, για παράδειγμα, στα αριστερά, στην πρώτη στήλη τα κοράλια της, ε, στα ζεστά έδατα. Αλλά ποια είναι η θετική είδηση από αυτή την έκθεση. Αν καταφέρουμε να διατηρήσουμε την θέρμανση του πλανήτη στον 1,5 βαθμό, όπως δηλαδή έχει τεθεί ως ο στόχος στην Συμφωνία των Παρισιών, θα είμαστε σε θέση να διατηρήσουμε σχεδόν όλα τα άλλα οικοσυστήματα και περισσότερα από αυτά σε, σε ζώνες εκτός ε, ιδιαίτερα υψηλού ε, κινδύνου. Για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά τα, τις περιοχές με τα φύκια, παρότι βέβαια θα επηρεάζεται η έκτασή τους, δεν θα είναι τόσο σοβαρές οι επιπτώσεις. Σε ό,τι αφορά, για παράδειγμα, από τις ε, παράκτης ε, περιοχές, ε, mangroves και άλλα είδη υγροτόπων, τα οποία δεν θα υποστούν τόσο σημαντικέ συνέπειε αν τελικά υπάρξει απόλυτη πολιτική δέσμευση για να παραμείνει η θέρμανση του πλανήτη σε επίπεδα κάτω των 2 ή κάτω του 1,5 βαθμού Κελσίου. Τώρα σε ό,τι αφορά την οξύνηση του ωκεανών θα πρέπει να πούμε ότι δεν έχουμε να κάνουμε μόνο με αυτήν την ε, πρόκληση δηλαδή τη οξύνηση, αλλά τον συνδυασμό αυτών των προκλήσεων δηλαδή τη θέρμανσης του πλανήτη σε συνδυασμό με την οξύνηση. Και βλέπετε ότι εάν έχουμε συνδυασμό της ε, ε, οξύνησης των ωκεανών με την θέρμανση του πλανήτη ακόμα πιο σοβαρές οι συνέπειες. Και γύρω στον 1,5 βαθμό βρισκόμαστε ακριβώς στη ζώνη όπου περνάμε από, την, ε, από τον μέτριο αν θέλετε κίνδυνο στον υψηλό κίνδυνο. Και φυσικά βέβαια τα επίπεδα κινδύνου είναι πολύ υψηλότερα αν έχουμε το σενάριο των 2 ε, βαθμών Κελσίου. Ακριβώς επειδή θα υπάρξουν αυτές οι φυσικοχημικές ε, επιπτώσεις και δράσεις. Τώρα τι συμβαίνει. Αυτό για την κατάσταση του πλανήτη, ότι δηλαδή ε, περνάμε σε μια πιο ασταθή περιοχή, ε, η φάση από πλευράς θερμοκρασίας μετά από μια σχετική σταθερότητα 5-6 χιλιάδων ετών και αυτό επηρεάζει δηλαδή και τις ε, χερσαίες περιοχές στις οποίες διαβιβούν ε, οι άνθρωποι. Οπότε σε ορισμένες ε, περιοχές ουσιαστικά οι θερμοκρασίες γίνονται απαγορευτικές για τη διατήρηση των, της ζωής σε αυτές. Και σε αυτό το γράφημα βλέπετε ακριβώς ποια είναι τα, ποιο είναι το εύρος των θερμοκρασιών ε, στο οποίο είναι δυνατόν να υπάρξει ανθρώπινη ζωή. Άρα δηλαδή η αύξηση του διοξιδίου του άνθρακα και η μείωση του οξυγόνου θα επηρεάσουν την ε, κατανομή, την βιοκατανομή στον πλανήτη. Και βλέπουμε για παράδειγμα στο δεύτερο διάγραφημα ότι έχουμε μια περισσότερη ε, επέκταση αν θέλετε της κατανομής ε, των ειδών ε, σε ψυχρότερες περιοχές και μείωση της κατανομής των ειδών στις θερμότερες περιοχές, δηλαδή επηρεάζονται και περισσότερο οι πολικές περιοχές. Με άλλα λόγια δηλαδή οι οργανισμοί αναγκάζονται να παραμένουν στα, στο εύρος θερμοκρασίας στο οποίο έχουν προσαρμοστεί. Δηλαδή με την κλιματική αλλαγή δεν βλέπουμε να υπάρχει μια αντίστοιχη προσαρμογή των, ε, της ζωής στην, ε, στις νέες Σε Τουλάχιστον δεν έχουμε παρατηρήσει κάτι τέτοιο. Αυτό σημαίνει με τη σειρά του μείωση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας. Και βλέπουμε δηλαδή το RCP 4.5 και το RCP 8.5 δηλαδή το ποια είναι η, εξέλιξη με βάση και πάλι δηλαδή τον, ε, το σενάριο του 1,5 ε, βαθμού και βλέπουμε το, ε, την, την μείωση της ε, και σε σίγουρα στα χαμηλότερα γεωγραφικά πλάτη έχουμε ακόμα πιο σοβαρή κατάσταση και παρατηρούμε δηλαδή ότι κάτι αντίστοιχο είχε συμβεί και κατά στις ε, προηγούμενες ε, περιόδους ε, προϊστορικά όπου είχαμε μεγάλη εξόντωση πάρα ειδών και πάλι δηλαδή αυτό είχε συμβεί κατά κύριο λόγο στα χαμηλότερα γεωγραφικά πλάτη. Άρα λοιπόν σε ό,τι αφορά την αλλαγή της κατανομής των ειδών υπάρχει ουσιαστικά δηλαδή μία αλλαγή και της ή παραγωγή τη βιομάζας, πράγμα το οποίο σχετίζεται ακριβώ με την οξύνηση των ωκεανών, με την υψηλότερη θερμοκρασία συγκεκριμένων περιοχών όπω ειδικότερα τη ακτική. Όπω βλέπετε και αν δείτε εδώ ε, στο σενάριο όπου δεν έχουμε μείωση των εκπομπών, σε καφέ χρόνο βλέπουμε πόσο μειώνεται η παραγωγή της βιομάζας ε, σε όλα τα γεωγραφικά πλάτη εδώ. Και μόνο αλλαγή, δηλαδή προς ε, αύξηση της ε, βιομάζας έχουμε μόνο κοντά στις πολιτικές περιοχές. Και στη, στη, στη, θαλάσσια ζωή έχουμε αντίστοιχη εξέλιξη, δηλαδή παρότι έχουμε αύξηση της βιομάζας σε ορισμένες περιοχές, στην, στην, στην πλειοψηφία έχουμε μείωση της βιομάζας, πράγμα το οποίο αντικατοπτρίζεται και στις δυνατότητες αλληλείας, όπως βλέπουμε δηλαδή στα, ε, στην τελευταία σειρά γραφημάτων. Αν δούμε λοιπόν, λίγο πιο προσεκτικά αυτή την κατάσταση θα διαπιστώσουμε ότι η σημερινή κατάσταση αποτελεί ακριβώς μια μεταβατική περίοδο προς αυτή την κατάσταση, ότι ήδη δηλαδή υπάρχει μείωση ε, των δυνατοτήτων της αλληλείας, υπάρχει ήδη ανακατανομή ε, των αποθεμάτων των ηχθείων και της θαλάσσιας ζωής και βλέπουμε στα περισσότερα γεωγραφικά πλάτη μείωση της ε, βιοποικιλότητας. Ε, ενώ σε κάποιες περιοχές, ειδικότερα δηλαδή στις πολιτικές, βλέπουμε να υπάρξει αύξηση, μια κάποια αύξηση της παραγωγικότητας της αλίας. Και παρότι συνεχίζεται μέχρι σήμερα αυτή η αύξηση στις πολιτικές ε, περιοχές μπορεί να είναι μόνο ένα παροδικό φαινόμενο ως αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής. Βέβαια, τα όσα αναφέρει αυτή η έκθεση και τα όσα περιλαμβάνουμε ως δεδομένα είναι προσωρινά δεδομένα γιατί δεν λαμβάνουμε υπόψη μας πλήρως τον περίπλοκο χαρακτήρα γιατί υπάρχει δηλαδή αλληλεπικάλυψη μεταξύ των διαφορετικών ειδών όπως ε, κατανέμονται και επηρεάζονται από τα επίπεδα διοξιδίου του άνθρακα και της υποξέες. Οπότε είναι σημαντικό να ληφθεί και αυτό υπόψη. Και ενώ στα δεξιά βλέπουμε ότι το εύρος της θερμοκρασίας και εξειδίκευση εξαρτάται από την ε, ηλικία των ε, ζώων. Δηλαδή, τα αυγά, για παράδειγμα, ή ε, τα ψάρια τα οποία βρίσκονται αναπαραγωγική ηλικία, είναι ιδιαίτερα ευάλωτα και είναι πολύ εξειδικευμένα σε ό,τι αφορά τη θερμοκρασία στην οποία μπορούν να επιβιώσουν. Αυτά λοιπόν τα ζητήματα, αυτέ οι διαφοροποιήσει, αν θέλετε, δεν λαμβάνονται υπόψη στα διάφορα δεδομένα τα οποία έχουμε συλλέξει για την έκθεση σε ό,τι αφορά ε, την, ε, το εύρο, για παράδειγμα, θερμοκρασία με βάση τι μελέτε που κάνουμε επιτόπια. Εδώ βλέπετε κάποια πρόσφατα δεδομένα τα οποία δεν έχουν ακόμα ληφθεί υπόψη στην ε, έκθεση, αλλά είναι σημαντικά γιατί καταδεικνύουν ακριβώ τι συμβαίνει σε ό,τι αφορά για παράδειγμα τον, ε, τη μάζα των ε, αυγών ε, σε ό,τι αφορά το γάτο του Ατλαντικού και τον ε, πολικό γάδο και βλέπουμε πώς υπάρχει άμεση επίπτωση της συμπληρωματικής οξύνησης των ωκεανών. Και αυτό βέβαια έχει με τη σειρά του επιπτώσει σε ό,τι αφορά την καταλληλότητα για αναπαραγωγή ε, αυτών των ειδών γάδου. Αριστερά δηλαδή για τον γάδο του Ατλαντικού και δεξιά για τον γάδο τον Αρκτικό. Βλέπουμε λοιπόν ότι τα, ε, ο, ο γάδος ε, του, ε, ο πολικός έχει προσαρμοστεί σε πολύ συγκεκριμένε θερμοκρασίε, γύρω στου 3 βαθμού, ενώ ο γάδο του Ατλαντικού είναι προσαρμοσμένο ή μπορεί να αναπαραχθεί σε μεγαλύτερο έυρος θερμοκρασία. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί βλέπουμε, για παράδειγμα, και πάλι εδώ με καφέ χρώμα την μείωση ε, της ε, καταλληλότητας ε, της, των περιοχών για αναπαραγωγή και πόσο δηλαδή ήδη μειώνονται οι δυνατότητες αναπαραγωγής σε ό,τι αφορά τις περιοχές που μπορεί να το πράξει ο ακτικός γάδος. Αυτό λοιπόν με τη σειρά του έχει τις δικές του επιπτώσεις στην παραγωγικότητα αυτών των αποθεμάτων. σίγουρα ακόμα και με την εφαρμογή της Συμφωνίας των ε, Παρισίων θα δούμε να λαμβάνουν χώρα οι ίδιες τάσεις αλλά όχι σε τόσο μεγάλο βαθμό. Παρόλα όμως ε, αυτά θα λάβει η χώρα δηλαδή μείωση της μάζας των ε, αυγών, μείωση των, της έκτασης των περιοχών αναπαραγωγής και ούτω καθεξής. Πώς μπορούμε λοιπόν να συνοψίσουμε ότι η ζωή γενικότερα είναι εξειδικευμένη σε ό,τι αφορά πολύ συγκεκριμένα εύρη θερμοκρασία. Ε, και οι αλλαγέ στον ωκεανό οδηγούν και σε μεταβολέ σε ό,τι αφορά τα αποθέματα των νυχθείων. Υπάρχει δηλαδή μείωση γενικευμένη των αποθεμάτων και ενώ σε κάποιε περιοχέ θα έχουμε μείωση αυτών των νυχθείων αποθεμάτων, σε άλλε θα έχουμε αύξηση, αλλά μπορεί να είναι παροδική. Και οι κοινότητε θα οι οποίες εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από αυτήν την ε, πηγή διατροφής θα έχουν ε, να αντιμετωπίσουν ζητήματα διατροφικής υγείας και ασφάλειας ε, της διατροφικής αλυσίδας και θα πρέπει να μειωθούν οι περαιτέρω πιέσει που δέχονται αυτά τα οικοσυστήματα, όπω για παράδειγμα η μόλυνση. Εάν υπάρχουν στα κατάλληλα πλαίσια πολιτική σε ό,τι αφορά τη διαχείριση τη αλληλεία θα έχουν θετικέ επιπτώσει στου ε, ανθρώπου και στα ηχθιαποθέματα. Βέβαια, δεν μπορούμε να κάνουμε λόγο για κλιματική αλλαγή χωρί να αναφερθούμε στην άνοδο τη στάθμη ε, ε, τη θάλασσα. Γιατί όλα αυτά τα ζητήματα και δηλαδή η αύξηση τη άνοδο τη της τη θάλασσα έχουν επιπτώσεις και σε ό,τι αφορά την αναπαραγωγικότητα των ηχθείων. Εδώ βλέπουμε για παράδειγμα την μείωση των στρωμάτων πάγου στην Γρυλανδία με βάση τα διαφορετικά σενάρια και βλέπετε ε, μια ε, πρόβλεψη έως ε, το 2300. Οπότε, σε ό,τι αφορά ε, τις προβλέψεις έως τα τέλη του αιώνα, έχουν αυξηθεί οι τάσεις οι οποίες προβλέπονται και κανείς δεν μπορεί να μας εγγυηθεί ότι θα παραμείνουν ίδιες οι, αυτές οι προβλέψεις γιατί δεν είμαστε ακόμα σίγουροι σε ό,τι αφορά που υπάρχουν συγκεκριμένα ορόσημα, θέλετε, δηλαδή σημαία καμπή σε ό,τι αφορά τις ε, περιοχές δηλαδή στρωματοπάγου. Και με την συνέχιση, για παράδειγμα, των, ε, της αξιοποίησης των ορυκτών καυσίμων, θα μπορούσαμε να οδηγηθούμε δηλαδή σε μια κατάσταση όπου θα ξεκινήσει μια ένα λιώσιμο αυτών των στρωμάτων πάγου χωρίς να μπορούμε να το σταματήσουμε με καταστροφικές συνέπειες. Βλέπουμε λοιπόν τα διαφορετικά, ε, τα διαφορετικά σενάρια ε, σε ό,τι αφορά δηλαδή τη σταθεροποίηση των ε, εκπομπών ή όχι για τις κλιματικές αλλαγές κατά 1,5 βαθμό και το πόσο δηλαδή μπορεί να επηρεαστεί το λιώσιμο των στρωμάτων πάγου με αντίστοιχη αύξηση της, ανώδου, και της, της στάθμης της Τι αυτό σημαίνει με τη σειρά του ότι μπορούμε να έχουμε περιπτώσεις αύξησης δηλαδή των, ε, της στάθμης ένα φαινόμενο το οποίο συνέβαινε για παράδειγμα ιστορικά μία φορά τον ε, κάθε αιώνα θα μπορούσε να είναι ένα ε, φαινόμενο το οποίο θα λαμβάνει χώρα πολύ πιο συχνά μέσα στις επόμενες δεκαετίες. Άρα λοιπόν συνοπτικά θα πρέπει να πούμε ότι 680 εκατομμύρια άνθρωποι διαβιούν σε παράκτητες περιοχές και 65 εκατομμύρια σε ε, κράτη μικρών ε, νησιών και κατά τον 20ο αιώνα ήδη ε, η στάθμη της θάλασσας αυξήθηκε κατά 15 εκατοστά. Τώρα, τη σήμερα ημέρα, η στάθμη της θάλασσας ανεβαίνει με διπλάσιους ρυθμούς και θα έχει φτάσει στο 1 μέτρο και 10 εκατοστά στο 2100 ή περισσότερα μέτρα στο 2300 αν δεν υπάρξει πολύ σαφής μείωση των εκπομπών. Και αυτό σημαίνει ότι θα υπάρξουν ε, πολύ σημαντικά καιρικά φαινόμενα, δηλαδή πολύ μεγάλος κίνδυνος ε, πλημμύρων και μείωση γενικότερα των χεσαίων εδαφών στο το 2050, αν δεν υπάρξει αντίστοιχη προσαρμογή. Δηλαδή, ορισμένα από αυτά τα κράτη, τα νησιωτικά κράτη, ενδεχομένως να εξαφωνιστούν τελείως. Υπάρχουν τώρα κάποια μέτρα προσαρμογής τα οποία μπορούν να εφαρμοστούν και σε ό,τι αφορά το ζήτημα της ε, αλληλεία. Ε, για παράδειγμα, ε, αν δεν υπάρξει καμία ανάληψη δράση, δεν θα υπάρξει καμία αλλαγή. Μπορεί να υπάρξει κατασκευή συγκεκριμένων αναχωμάτων για την προστασία παράκτιων περιοχών διατηρώντας και, τα, και τις σχετικές περιοχές αναπαραγωγής για τους εχθείς μπορεί να υπάρξει μια άλλη ε, προσαρμογή, δηλαδή με την αύξηση ουσιαστικά του ύψους στο οποίο κατασκευάζονται οι οικισμοί ή για παράδειγμα μπορεί να υπάρξει αναχωμάτωση ε, κοντά, στην, ε, κοντά στις ακτές όπως γίνεται για παράδειγμα στην, και στη Γερμανία αλλά και στις χατοχώρες ιστορικά για την προστασία δηλαδή των νησιωτικών περιοχών ή μπορεί να υπάρξει μετακίνηση Πράγμα το οποίο, δηλαδή αυτή η μετακίνηση ε, των ε, οικισμών θα μπορούσε να είναι ε, κάτι το πιο θετικό σε ό,τι αφορά τα οικοσυστήματα. Υπάρχουν λοιπόν μια σειρά από διαφορετικέ εναλλακτικέ οι οποίε έχουν εξεταστεί και μια ακόμα φορά κάναμε εδώ την, μια αξιολόγηση κινδύνου λαμβάνοντα υπόψη τι δυνατότητε ακριβώ που μα παρέχουν αυτέ οι διαφορετικέ δυνατότητε προσαρμογή και βλέπουμε εδώ μια σύγκριση μεταξύ του, δηλαδή καμία προσαρμογή στα αριστερά και στα, στην, δεξιότερη στήλη τεράστια προσαρμογή. Βλέπουμε όμως ε, πως ε, εάν υπάρχουν, μιλάμε για πόλεις οι οποίες έχουν και αρκετούς πόρους στη διάθεσή τους μπορούν να παραμείνουν σε χαμηλά επίπεδα κινδύνου ενώ άλλες ε, μικρότερες κοινότητες θα βρίσκονται πολύ κοντά στις, στα όρια της μετακίνησής τους, αν προσαρμογής τους ειδικότερα τις ε, περιοχές χαμηλού υψομέτρου, όπου θα υπάρχουν δηλαδή πολύ περιορισμένες δυνατότητες σε ό,τι αφορά την ε, προσαρμογή. Άρα λοιπόν ε, πρέπει να κάνουμε λόγο για προσαρμογή εφόσον υπάρχει τέτοια δυνατότητα. Θα υπάρξουν πάντω περιορισμοί σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα προσαρμογή και αυτό θα επηρεάσει ειδικότερα τι ε, κοινότητε ε, που βασίζονται στην Αλία. Υπάρχουν εδώ και κάποιες άλλες προκλήσεις που αφορούν ε, κοινωνικά θέματα. Θα πρέπει καταρχήν να βρούμε τις πιο ευάλωτες ομάδες ανθρώπων, αυτούς που θα πληγούν περισσότερο, αυτούς που δεν έχουν δυνατότητα αντιμετώπισης. Αλλά βεβαίως οι συνέπειες όσον αφορά την κλιματική αλλαγή θα πρέπει να τις δούμε διότι έχουν πολύ μεγαλύτερη διάρκεια στο χρόνο σε σχέση με θέματα διακυβέρνησης. Υπάρχει κατακαιρματισμός όσον αφορά την αντιμετώπιση της, ε, από άποψη διακυβέρνησης. Βεβαίως εδώ δεν υπάρχει μια ενιαία αντιμετώπιση και απάντηση και θα πρέπει εδώ να υπάρξει μια διαβούλευση και μια εμπειρογνωμοσύνη όσον αφορά τη γενικότερη αντιμετώπιση θεμάτων που αφορούν τους ωκεανούς και που ξεπερνούν ε, τις ε, εθνικές αρχές. Βλέπουμε ότι πολλές φορές οι απαντήσεις δεν είναι αρκετά ε, αποτελεσματικές, ιδιαίτερα όσον αφορά την αντιμετώπιση αυτών των σημαντικών αλλαγών και πληγμάτων που προκαλούνται σε παράκτιες περιοχές. Επίσης το κόστος τους πιστεύω δεν έχει εκτιμηθεί ακόμα σωστά. Λύσεις που μπορεί να βρεθούν, προσαρμογές σε σχέση με τα οικοσυστήματα, ποιες είναι οι περιοχές αυτές οι οποίες θα πρέπει να προστατευθούν κατά προτεραιότητα και βεβαίως ε, οι δυνατότητες να επιλεγεί μία ή άλλη εναλλακτική λύση ανάλογα με τις ε, προστατευόμενες ε, περιοχές, ε, οικοσυστήματα που πρέπει να προστατευθούν, δυνατότητες δημιουργίας αναχωμάτων είτε μετατόπισης κάποιων συγκεκριμένων πληθυσμών. Όλα αυτά τα μέτρα δεν μπορεί να είναι αποτελεσματικά παρά μόνο εάν εφαρμοστεί σωστά και ολοσχερός η Συμφωνία του Παρισιού το θέμα τώρα της υπερεκμετάλλευσης των αλληλευτικών αποθεμάτων σε κάποιες περιοχές και βεβαίως ε, οι αρνητικές επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος ε, καθώς και η μη τήρηση κάποιων οικονομικών περιορισμών. Θαλάσσιες περιοχές που προστατεύονται, η εκμετάλλευση των αλληλευτικών αποθεμάτων και η τήρηση ε, των περιορισμών. Ολοκληρώνω. Η έκθεση αυτή καλύπτει το 80% της επιφάνειας του πλανήτη. Προσπαθεί να αντιμετωπίσει με τρόπο ολοκληρωμένο όλες αυτές τις επιπτώσεις, οι οποίες μπορεί να συνεχιστούν για τις επόμενες γενιές, αλλά μπορεί να αντιμετωπιστούν και να εξουδετερωθούν, να μετριαστούν. Χρειάζεται συντονισμένη δράση, διότι πρόκειται για αλλαγές οι οποίες ε, αποτελούν απειλές για όλους τους ωκεανούς. Πρόκειται για μέτρα τα οποία θα πρέπει να ληφθούν με έναν αποτελεσματικό και ολοκληρωμένο τρόπο και θα πρέπει σε κάθε περίπτωση η επιστημονική δράση, η γνώση, η εμπειρογνωμοσύνη καθώς και η κατάρτιση των τοπικών κοινωνιών, η ευαισθητοποίηση να αντιμετωπίσουν αυτό που σήμερα με κατακαιρματισμένο τρόπο αντιμετωπίζεται από τις τοπικές κοινωνίες. Χρειάζεται η επιστημονική γνώση να γίνει αποδεκτή και ίσως όλοι εμείς, όλοι εμείς σε ένα μεγάλο βαθμό θα πρέπει να ευαισθητοποιηθούμε για να συνεισφέρουμε. Τώρα, όσον αφορά την υλοποίηση όλων αυτών των μέτρων και των προτάσεων. Έχουμε την ε, έκθεση που αντιμετωπίζει την υπερθέρμανση του πλανήτη, τι μπορούμε να κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε την αύξηση της θερμοκρατίας, τα μέτρα που έχουν ε, προταθεί, οι νέες τεχνολογίες για να στηρίξουν αυτήν την αντιμετώπιση της αύξησης ε, της θερμοκρασίας, μέτρα προσαρμογής και κατεύθυνση νέων μέτρων οικονομικών. Τέλος της ε, εκμετάλλευσης σε κάποια μη εκμεταλλευόμενα σήμερα κοιτάσματα, παραδείγματο χάρη ε, φυσικού αερίου και πετρελαίου. Η έκθεση 1.5 η οποία περιέχει συγκεκριμένα μέτρα για τη μετατροπή της πολιτικής μας θα πρέπει να αποτελέσει μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις. Ολοκληρώνω κοιτώντας αυτές τις τρεις εκθέσεις και τα μηνύματά τους που είναι η αντιμετώπιση της ε, αύξησης της θερμοκρασίας, θέματα που κάθε χρόνο επανέρχονται, θέματα που αφορούν τους ωκεανούς, Κάθε επιλογή μετράει, κάθε επιλογή έχει τα αποτελέσματα και συνεισφέρει και πρόκειται για πολιτικά, κοινωνικά θέματα, τα οποία μας αφορούν όλους, όπως εξάλλου υπογραμμίζουμε στην έκθεση αυτή και στα πορίσματα του συνεδρίου που χώρα στην Ορδηγία τον προηγούμενο μήνα. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Thank you, Professor, for trying to finish on a positive note. Ευχαριστούμε κύριε καθηγητέ, διότι τουλάχιστον τελειώσαμε με ένα πολύ θετικό μήνυμα. Τι έχετε να πείτε συνολικά για τις εκπομπές, αυξάνονται ή μειώνονται. Κοιτάξτε, δεν έχουμε ακόμα φτάσει στο υψηλότερο βαθμό των εκπομπών. Πιστεύω ότι συνεχίζονται σε γενικό, γενικές μετρήσεις. Κάποιες χώρες δεν έχουν φτάσει ακόμα τον βαθμό εκπομπών. Η Επιτροπή έχει ζητήσει το λόγο πριν πάνω το λόγο τα μέλη της Επιτροπής Αλίας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πρόεδρε. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που σήμερα ξεκινάει αυτή η συζήτηση εδώ στην Επιτροπή Αλίας. Θέλουμε να συγχαρούμε την Διακυβερνητική Επιτροπή, τον εισηγητή, τον κύριο Πέλτνερ, για την παρουσίαση αυτή. Νομίζω ότι όλοι θα συμφωνήσετε ότι πρέπει για μια ανησυχητική κατάσταση και θεωρώ ότι εδώ η Επιτροπή Αλίας είναι το κατάλληλο όργανο για να συζητήσει τα θέματα αυτά. Βεβαίω πρόκειται για την πιο σημαντική πρόκληση του αιώνα μας η αύξηση της θερμοκρασίας, κάτι που αναγνωρίστηκε και από τη Συμφωνία του Παρισιού. Είναι κάτι που σαφώς και όλοι έχουμε συνειδητοποιήσει. Ο ρόλος των ωκεανών όσον αφορά τη ρύθμιση του κλίματος οι ωκεανοί μα βρίσκονται στην πρώτη γραμμή μια εξαιρετικά επίγουσας κατάσταση που μας απασχολεί και μας απειλεί όλου. και θα πρέπει να δούμε ποιε είναι οι επιλογέ μα, οι οποίε θα είναι καθοριστικέ για το μέλλον των ωκεανών και για το μέλλον τη ανθρωπότητα. Αυτή η έκθεση μας δίνει πολύ σημαντικά στοιχεία και επιστημονικά δεδομένα βάσει των οποίων θα πρέπει να πάρουμε τις αποφάσεις μας. Γι' αυτό και είναι πάρα πολύ σημαντική είναι πολύ σημαντική καθότι η Προεδρία της Χιλής το 2020-2025 θέλει να δώσει ένα καθοριστικό ρόλο όταν πάρουν τις αποφάσεις τους το Δεκέμβριο του 2020 θεωρούμε ότι ακριβώς επειδή η Προεδρία της Χιλής έχει εντοπίσει σαν μία από τις προεδριότητες της, ε, τους ωκεανούς, θα πρέπει και η επόμενη συνεδρίαση της ε, ΚΑΠ 21 να λάβει υπόψη της ακριβώς το ρόλο των κενών. Όπως εξάλλου ε, βλέπουμε και στις ε, προτεραιότητες της Συμφωνίας των Παρισιού. Ποια είναι τα μέτρα αυτά που θα πρέπει να ληφθούν για να μετριαστούν ε, οι επιπτώσεις ε, της αλλαγής του κλίματος ε, επί των ωκεανών. Πώς μπορούμε να προστατεύσουμε τα θαλάσσια οικοσυστήματα. Πρόκειται για εξαιρετικά σημαντικές προκλήσεις για τις κυβερνήσεις, για την αλία. Είδαμε ότι υπάρχει σήμερα μεγάλη μεταβολή όσον αφορά τα είδη των αλλιευμάτων, τις περιοχές στις οποίες βρίσκονται. Πρόκειται για προκλήσεις όσον αφορά τη διαχείριση και σε τοπικό επίπεδο των αλλιευμάτων, αλλά και για τις νέες διαπραγματεύσεις και συζητήσεις μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών, ιδιαίτερα για τις αναψώμενες χώρες. Οι οργανισμοί που παίζουν ρόλο καθορισμού και διαχείρισης των αλλιευμάτων στον τομέα αυτό, θα πρέπει να κοιτάξουν ιδιαίτερα ποιε θα μπορούσε να είναι οι εναλλακτικέ. Γι' αυτό και είναι καθοριστική η έκθεση αυτή της Διακυβερνητικής Επιτροπής και οι εναλλακτικέ μας προτείνει. Νομίζω ότι τα επιστημονικά δεδομένα που διαθέτουμε σήμερα όσον αφορά τις επιπτώσεις στους ωκεανούς της αλλαγής του κλίματος είναι κάτι που θα παραμείνει στην, στις προτεραιότητές μας για τα επόμενα χρόνια. Η κλιματική αλλαγή είναι μία από τις σημαντικές προτεραιότητες, όπως εξάλλου η Ούρσουλα Leyen έχει ανακοινώσει. Μία από τις προτεραιότητες αυτής της Επιτροπής θα είναι και οι ωκεανοί. Θα πρέπει να παραμείνουμε ενεργοί στην δράση μας και νομίζω ότι εδώ θα πρέπει όλοι μαζί να συγκεντρωθούμε και να συνεργαστούμε στην αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου. Ε, Σα ευχαριστώ κύριε καθηγητά για την παρουσίασή σας, παρουσίαση αυτού του σημαντικού ε, εγγράφου όσον αφορά την κλιματική αλλαγή. Είναι σαφές ότι η κλιματική αλλαγή έχει πολύ μεγάλη επίδραση στους ωκεανούς, υπερθερμάνση των υδάτων, λιγότερο οξυγόνο, λιγότερα, περισσότερα ε, οξέα και αυτό βεβαίως έχει μεγάλο, μεγάλη επίδραση ε, στα αλλιευτικά αποθέματα, τη δυνατότητα αναπαραγωγής κλπ και βεβαίως ε, ε, επηρεάζεται ε, και το πλήθος των αλλιευμάτων καθώς επίσης και η σύσταση των ιδίων. Αλλά σε σχέση με την αλληλεία και σε σχέση με εμά εδώ στην Ευρώπη νομίζω ότι εμείς έχουμε ήδη δημιουργήσει ένα σύστημα βιώσιμης αλληλεία που βασίζεται βεβαίως ε, στις ε, αλλιευτικές ε, ποσοστώσεις καθώς επίσης και στην ανάπτυξη πολιτικών που λαμβάνουν υπόψη τις, τους επιστήμονες και τα όσα λένε για την ε, κλιματική αλλαγή. Επίσης, εμείς εφαρμόζουμε την αρχή της πρόληψης. Ε, είδαμε και πριν πόσο σημαντική είναι η αρχή της πρόληψης, την οποία εμείς εφαρμόζουμε στην Αλία σε γενικές γραμμές ε, έχει βελτιωθεί η κατάσταση των αποθεμάτων, των αλλιευτικών αποθεμάτων που υφίστανται, διέπονται από, του, από τις ποσοστώσεις. Επίσης ε, ε, γίνεται λόγος για τον βακαλάο της ε, Βαλτικής που δεν είναι θέμα υπεραλίευσης αλλά είναι θέμα έλλειψης αναπαραγωγής. Πιστεύουμε ότι η αλληλεία η οποία είναι μια σημαντική οικονομική δραστηριότητα έχει υποφέρει από την, και υποφέρει από την κλιματική αλλαγή. Μιλισμονούμε ότι η αλληλεία είναι μια σημαντική οικονομική δραστηριότητα η οποία ακριβώς υφίσταται τις επιπτώσεις και είναι θύμα επομένως της κλιματικής αλλαγής. Ήθελα να πω και κάτι άλλο σε σχέση με τα ε, ψάρια. Τα ψάρια είναι μια σημαντική πηγή πρωτεΐνης ε, και ε, ξέρετε ότι το αποτύπωμα του, της είναι χαμηλότερο από οποιαδήποτε άλλη εξορυκτική ε, δραστηριότητα. Ε, θα ήθελα να τελειώσω λέγοντας ότι βεβαίως εμείς θέλουμε να αγωνιστούμε και εμείς κατά αυτής της ε, τεράστιας απειλής γιατί μας ενδιαφέρει και η επιβίωση της αλληλείας καθώς επίσης και των αλληλευτικών αποθεμάτων. Ευχαριστώ πολύ κυρία Αγγιλάρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Αναμφίβολα τα όσα ακούσαμε είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα και σημαντικά και έγκαιρα μάλιστα. Στην ε, ε, πολιτική, για τη διαμόρφωση πολιτικών, πρέπει κανείς να λαμβάνει υπόψη ε, τις επιστημονικές εισηγήσεις. Και εδώ έχουμε μία σημαντική μια εξαιρετική εισήγηση. Εγώ αυτό που θα ήθελα να κάνω είναι το εξής, να υποβάλω συγκεκριμένα ερωτήματα Πρόκειται για θέματα τα οποία συζητούνται και ερευνώνται εδώ και πολλά χρόνια και θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στην μεταρρύθμιση της αλλιευτικής ε, ε, πολιτικής και χρειάζεται και ριζική με κάθε έννοια που μπορεί να έχει αυτό ο επιθετικός προσδιορισμός της αλλιευτικής πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πέρα από το σύστημα που ανέφερε ο κύριος Μηγιαμών, το σύστημα των ποσοστώσεων, ε, της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης κλπ. Έχουμε και επίσης μια άλλη σειρά μέτρων, ας πούμε, ε, έχουμε εγκρίνει κάποια σχέδια διαχείρισης ε, τα οποία θα πρέπει οπωσδήποτε να βελτιωθούν και να διευρυνθούν γιατί σε πολλές περιοχές όπως ας πούμε η Μεσόγειος ή ο Εύξηνος Πόντος θα πρέπει να, ε, διαχειρίζονται, να τα διαχειριζόμαστε βάσει των σχεδίων διαχείρισης ε, και οπωσδήποτε να βελτιωθεί η κατάσταση έτσι ώστε να διαχειριστούμε καλύτερα το σύνολο της καταστάσεως ε, και να λάβουμε υπόψη και τα όσα αποφασίστηκαν στην διάσκεψη των Παρισίων γιατί εμείς στην Ευρώπη είμαστε δεσμευμένοι απέναντι σε αυτά. Εμείς ε, ε, οπωσδήποτε ε, είμαστε υποχρεωμένοι άλλωστε να αποτελέσουμε παράδειγμα όσον αφορά την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Όμως, συγκεκριμένε ερωτήσεις στον κύριο καθηγητή. αυτά τα χρόνια, δεν είναι πάρα πολλά βέβαια, που τα σχέδια διαχείρισης έχουν αρχίσει να υλοποιούνται τα τελευταία δύο-τρία χρόνια. Είστε είστε της άποψης ότι αυτή η αλληλευτική πολιτική και όλα αυτά τα στοιχεία της ε, μέγιστης ε, βιώσιμης ε, απόδοσης κλπ. μπορούν να μας βοηθήσουν, να μας οδηγήσουν στην εκπλήρωση αυτών των στοιχείων ή θα πρέπει να πάρουμε και επιπλέον μέτρα. Είμαστε στο σωστό δρόμο γιατί και όσον αφορά τις ε, υποχρεώσεις εκφόρτωσης που ήταν μια δύσκολη κατάσταση και δημιουργεί πολλά προβλήματα. Πιστεύετε ότι είμαστε στο σωστό δρόμο ή θα πρέπει να πάρουμε και επιπλέον μέτρα τα επόμενα χρόνια. Well, uh, Πρόεδρος, αναφερθήκατε ε, στην ανάγκη ανασύστασης ε, των προβληματικών αλλιευτικών αποθεμάτων και στην ε, Επιτροπή Περιβάλλοντος ε, θίξαμε το θέμα ε, των αποδεκατισμένων αλλιευτικών αποθεμάτων. Μπορούμε να επανασυστήσουμε αυτά τα προβληματικά αποθέματα μέσω και της απαγόρευσης αλίευσης έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή. Απάντηση. Οπωσδήποτε αυτό εξαρτάται από τα συγκεκριμένα είδη καθώς επίσης ε, και την επιτρεπόμενη αλίευση, αλλά οπωσδήποτε ε, η κλιματική αλλαγή αποτελεί μια επιπλέον, έναν επιπλέον ε, παράγοντα πίεσης ε, της, ε, που οδηγεί στη μείωση των αποθεμάτων. Η απαγόρευση ή η μείωση της, του επιτρεπόμενου αλλιεύματος βεβαίως είναι ένα καλό πρώτο βήμα. Ε, πρέπει να υπογραμμιστεί ότι τα οικοσυστήματα στα οποία αλλιεύεται αποτελούν ακριβώς τον, τον χώρο στον οποίο ζουν και αναπαράγονται τα αλλιεύματα. Έχουμε προβλήματα ας πούμε με τον γάδο, τα, αποθέματα του γάδου της ε, ε, Βαλτικής και οι κακές περιβαλλοντικές συνθήκες αυτές τις ε, περιοχές έχουν δημιουργήσει επιπλέον επιβαλλοντικούς παράγοντες. Ε, και επομένως ε, και λόγω της έλλειψης οξυγόνου και λόγω της κλιματικής αλλαγής υπερθέρμανσης των υδάτων ε, πιέζεται ακόμα περισσότερο ο γάδος της Βαλτικής και της Βόρειας θάλασσης. Οπωσδήποτε είναι μια κατάσταση που παρουσιάζει ιδιαίτερες δυσκολίες αλλά πάντα ένα πρώτο βήμα είναι καλό και η απαγόρευση αλίευσης μπορεί να είναι ένα πρώτο καλό βήμα. Όσον αφορά την σειρά συναντήσεων που είχαμε για την κατάσταση των ωκεανών, να σας πω το εξής, που το χρησιμοποιώ και σαν μήνυμα, το χρησιμοποίησα στα, στις διαφάνειές μου. Η δημιουργία δικτύων προστασίας, εκεί που η κατάσταση των αλλιευμάτων είναι ιδιαίτερος επικίνδυνη, ε, μπορεί να οδηγήσει σε μάλλον εξαρτάται από μια σειρά παραγόντων. Ε, δηλαδή, σε περιοχές οι οποίες ε, ε, αντιμετωπίζουν προβλήματα θα πρέπει και να προστατευτούν τα λεύματα στην ε, προστατευόμενη περιοχή και θα το επιτύχετε αυτό μέσω των συγκεκριμένων μέτρων αλλά και θα δημιουργήσετε παραπέρα περιοχές όπου μπορεί να συνεχιστεί η αλλιευτική δραστηριότητα η οποία κατανοούμε ότι πρόκειται για εργασία και για μια βιοποριστική δραστηριότητα. Το σημαντικό είναι να δημιουργηθεί δίκτυο προστατευόμενων ε, περιοχών στις παράκτιες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς επίσης και στους ωκεανούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί μόνο με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσετε ε, να δημιουργήσετε συνθήκες ε, ικανές μετανάστευσης των ψαριών σε άλλες προστατευόμενες περιοχές και ενδεχομένως και σε περιοχές όπου η αλίευση είναι λιγότερη. Ευχαριστώ πολύ, καθηγητά. Το συζητήσαμε αυτό στην Επιτροπή μας. Έχουμε πάρα πολλές τέτοιες προστατευόμενες ε, περιοχές. Ε, απάντησα, απαντήθηκε η ερώτησή σας. Η κυρία Αγγιλέρα. Θα ήθελα πιο συγκεκριμένα να ρωτήσω εάν βοηθά, αν βοηθάει η μείωση της ελευτικής δυνατότητας. Αυτό το ξέρουμε ε, ότι βοηθάει και το κάνουμε ήδη. Τα σχέδια διαχείρισης όμως, τα οποία έχουν ήδη αρχίσει να ε, υφίστανται και στα πλαίσια των οποίων ε, με τα συστήματα των ποσοστώσεων, των τάξ και τα λοιπά, μειώνεται η αλίευση για τη Μεσόγειο, ας πούμε, που ήταν το πρώτο σχέδιο διαχείρισης ε, και για τα βανθυπελαγικά ε, είδη για τα οποία θα υπάρχει μείωση του χρόνου της ελιευτικής προσπάθειας. Ρωτώ λοιπόν, όλα αυτά είναι ο σωστός δρόμος. Βεβαίως θα χρειαστούμε περισσότερα χρόνια έτσι ώστε να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε πραγματικά το αποτέλεσμα. Αλλά θεωρεί ε, ο κύριος καθηγητής ότι είναι ο σωστός δρόμος. Ε, γιατί με τα συστήματα των ποσοστώσεων, των RMS, ε, πηγαίνουμε προς το σωστό δρόμο ή δεν κάνουμε κάτι. Ε, γιατί είχα κάπως την εντύπωση ότι η άποψή του είναι ότι δεν είμαστε στο σωστό δρόμο ή δεν κάνουμε και πολλά πράγματα. Κοιτάξτε, υπάρχει αβεβαιότητα, αλλά έτσι και αλλιώ σε κάποιες περιοχές μπορεί να πρέπει να μειωθεί η αλλά σε γενικές γραμμές το πώς αντιδρούν τα αλλιεύματα, αν θέλετε, στην αλλαγή του κλίματος, εδώ υπάρχουν διάφορες παρατηρήσεις, υπάρχουν ε, διάφορες έρευνες ε, και παρατηρήσεις. Δεν αντιδρούν με τον ίδιο τρόπο όλα τα είδη ηχθείων στην αλλαγή του κλίματος και στην αύξηση της θερμοκρασίας. Υπάρχουν ε, λοιπόν ε, και συνεχίζονται όλες αυτές οι έρευνες και νομίζω ότι μόνο με παρατήρηση και με σύγκριση των αποτελεσμάτων ε, των επιστημονικών ερευνών μπορεί κάποιος να έχει μια τελική απάντηση. Η μείωση παντός της πίεσης επί των αλλιευμάτων, επί όλων των ειδών Σίγουρα εδώ είναι ένα από τα προβλήματα. Ο κύριος Σάλιβαν. Η κυρία Σάλιβαν, συγγνώμη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ στην Επιτροπή Ένβη αντιμετωπίσαμε και συζητήσαμε όλα αυτά τα αποτελέσματα αυτής της ε, έκθεσης, τα πορίσματα, τα οποία είναι πάρα πολύ ανησυχητικά και δημιουργούν ε, ερωτηματικά. Τι μπορούμε να κάνουμε για να αλλάξουμε τα πράγματα, η οποία φαίνεται να είναι καταστροφικά. Χαίρομαι γιατί αναφέρεστε στις προστατευόμενες περιοχές, αναφέρεστε και στις δυνατότητες που πρέπει να έχουμε να συνδυάσουμε τις ε, προστατευόμενες αυτές ε, περιοχές και να βρούμε τρόπους να αντιστρέψουμε την κατάσταση. Κύριε καθηγητά, άκουσα πολύ προσεκτικά αυτά που είπατε για τις περιοχές, για τα οικοσυστήματα, για τον τρόπο αναπαραγωγής αλλά όσον αφορά τα θέματα προστασίας ε, κάποιων άλλων οργανισμών όπως ε, του πλανκτών, οι επιπτώσεις επί αυτών των συστατικών των ωκεανών της αύξησης της θερμοκρασίας εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και επειδή θέλουμε να έχουμε έναν ηγετικό ρόλο στην προστασία των ωκεανών, τι μπορούμε να κάνουμε πολύ συγκεκριμένα για να διασφαλίσουμε ότι σε όλα τα επίπεδα κάνουμε κάτι για να μετριάσουμε τις αρνητικές επιπτώσεις αυτής της υπερθέρμανσης του πλανήτη επί των ωκεανών. Ευχαριστώ πολύ. Θα πάρουμε και άλλη ερώτηση. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον ε, καθηγητή για την παρουσίασή του και για τις εξηγήσεις που έδωσε μέχρι τώρα. Έχω την εντύπωση ότι είναι σημαντικό να υπογραμμίσουμε εδώ ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε όλες αυτές τις ε, περιοχές αλίας και ιδιαίτερα τη Βόρεια Θάλασσα με έναν βιώσιμο τρόπο. Υπάρχουν υποσωστώσεις ε, και θέλουμε όλη η δραστηριότητα της αλίας να γίνει βιώσιμη. Για κάποια αποθέματα έχουμε ήδη θετικά αποτελέσματα. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας στις μελλοντικές μας προσπάθειες ε, εκεί που τα αποτελέσματα είναι ήδη θετικά και στη Βόρεια Θάλασσα και αλλού. Στην έκθεσή σας βλέπουμε ότι στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εξάλλου το επανέλαβε αυτό και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είμαστε πάρα πολύ θερμοί υποστηρικτές αυτών των προσπασιών. Όμως υπάρχουν χώρες που θέλουν να πάρουν αυτή την έκθεση και να την πετάξουν στα σκουπίδια. Θα ήθελα να ξέρω ποιες είναι οι χώρες αυτές που αρνούνται ε, αγνοούν αυτά τα φαινόμενα και απορρίπτουν τα πορίσματά σας. Πριν ξεκινήσετε την παρουσίασή σας, μας δείξατε ένα μικρό βιντεάκι. Λέτε αλλάζουμε τον πλανήτη, τροποποιούμε τον πλανήτη. Αυτό είναι η πραγματικότητα. Υπάρχουν σήμερα κάποιοι που αρνούνται ότι υπάρχει κλιματική αλλαγή, λένε ότι τίποτα το περίεργο δεν συμβαίνει, πρόκειται για ένα φυσικό φαινόμενο. Υπάρχουν σήμερα άνθρωποι ε, στον πλανήτη, υπάρχει το ΖΙΕΚ, αλλά υπάρχουν και οι δικές σας μελέτες και έρευνες που θα πρέπει να ληφθούν πιο σοβαρά υπόψη. Και αναρωτιέμαι, γιατί σήμερα η κλιματική αλλαγή αντιμετωπίζετε με αυτό τον τρόπο. Εσείς, η έκθεσή σας, η οποία είναι αξιόλογη, εγώ είμαι πεπισμένος γι' αυτό, συνεχίζει να αντιμετωπίζεται σαν γελία από κάποιους και μάλιστα μέλη του Κοινοβουλίου μας. Όσον αφορά, παραδείγματο χάρη, την αύξηση της θερμοκρασίας ε, του νερού, των ωκεανών, η οποία συνεχίζει να συμβαίνει δύο ή τρεις βαθμοί επιπλέον είναι κάτι το οποίο θα συμβεί χωρίς να μπορούμε από ό,τι φαίνεται να το αποφύγουμε. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να το καταγράψουμε. Θεωρείτε ότι αυτό το φαινόμενο της αύξησης της θερμοκρασίας είναι κάτι που μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε, που μπορούμε να το ανατρέψουμε ή όχι.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 Ας ξεκινήσουμε με το πλακτόν. Βλέπουμε λοιπόν στι ίδιε ομάδε οργανισμών τα ίδια φαινόμενα με αυτέ που βλέπουμε στα αλεύματα. Δηλαδή, αρχίζει η μετακίνησή του σε διαφορετικό γεωγραφικό πλάτο. Ε, και ε, τα έργα θερμοκρασιών έχουν καταδείξει σημαντικά ότι πράγματι συγκεκριμένα δηλαδή ήδη είναι εξειδικευμένα σε συγκεκριμένα εύρη θερμοκρασία. Άρα λοιπόν η αλλαγή τη θερμοκρασία στον ωκεανό αρχίζει να αναμειγνύει διαφορετικά οικοσυστήματα, που σημαίνει θα υπάρξουν διαφορετικέ διατροφικέ αλυσίδε, διαφορετικά είδη τα οποία θα έρθουν σε επαφή μεταξύ του. Και έτσι όσο πιο μεγάλη θα είναι η αλλαγή τη θερμοκρασία στον ωκεανό που θα επιτρέψουμε να λάβει η χώρα, τόσο πιο μεγάλε θα είναι οι αλλαγέ που θα συμβούν στα οικοσυστήματα. Και νομίζω πω υπάρχει στην επιστημονική κοινότητα συνένεση ότι εάν κινηθούμε πάνω από 1,5 βαθμό θέρμανση δηλαδή του πλανήτου, περνάμε σε ένα τελείω διαφορετικό σενάριο, σε ένα τελείω διαφορετικό πλανήτη από αυτό που γνωρίζουμε. Και σε κάποιο βαθμό αυτό ισχύει και για τον τρόπο με τον οποίο θα αναπτυχθούν σε διαφορετικά πλέον σημεία διαφορετικά οικοσυστήματα. Ακριβώς δηλαδή λόγω ακριβώς αυτής της ε, μετακίνηση ε, του, του περάσματος σε μια εποχή με χαμηλότερη βιοπικιλότητα και λόγω της μετακίνησης των ειδών θα δούμε εντελώς νέα οικοσυστήματα. Σε ό,τι αφορά τώρα την μείωση των εκπομπών με βάση τη Συμφωνία των Παρισίων, πραγματικά δεν θα πρέπει να είναι αδιαπραγμάτευτο αυτό ο στόχο. Ελήφθη η σχετική απόφαση και τώρα ήρθε η στιγμή να εφαρμοστεί στην πράξη. Και γνωρίζετε ότι μπορούμε να κάνουμε πολλούς συμβιβασμούς γιατί εσείς ως αρμόδιοι για τη χάραξη της πολιτικής θα πρέπει να κάνετε πολλούς συμβιβασμούς αλλά θα πρέπει να ε, έχετε κατά νου ότι εδώ πρόκειται για κάτι το οποίο δεν είναι ευέλικτο. Δηλαδή δεν μπορείτε να παρεκκλίνετε από τις εκπομπές τις οποίες έχετε συμφωνήσει έτσι ώστε να διατηρηθεί η θέρμανση του πλανήτη στο έως και 1,5 βαθμό Κελσίου προκειμένου να διατηρηθεί η παραγωγικότητα και στους ωκεανούς και για, τα, για την αλληλεία και προκειμένου να αντισταθμίσουμε τις ε, ζημίες οι οποίες έχουν ήδη λάβει η χώρα με βάση την κλιματική αλλαγή. Γιατί και στη συνάντηση όσαν σε ωκεανοί μας υπήρξε μια έκθεση η οποία παρουσιάστηκε από τον ε, Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας ε, του ΦΑΟ σε ό,τι αφορά την παραγωγικότητα με βάση τις αλληλίες στον ωκεανό και εκεί καταδείχθηκε ότι εάν ε, παραμείνουμε εκεί που πρέπει σε ό,τι αφορά τους στόχους, ενδεχομένως να είναι δυνατό όχι μόνο να διατηρηθεί, αλλά και να αυξηθεί λίγο η παραγωγικότητα. Και επίσης θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονό ότι σε ό,τι αφορά τι παράκτητε περιοχέ ενδεχομένω να προκύψουν κάποιε νεκρέ ζώνε όπου δεν θα υπάρχει δηλαδή ε, δεν υπάρχει δυνατότητα να διατηρηθεί ζωντανό οργανισμό και κατά συνέπεια ούτε και υδατοκαλλιέργεια. Οπότε ε, το ζητούμενο εδώ είναι να δημιουργήσουμε ένα σύστημα το οποίο θα είναι απόλυτα βιώσιμο και ποιε θα είναι οι ιδιότητε ενό τέτοιου συστήματο. Ποιε δηλαδή θα είναι οι παράμετροι τι οποίε θα πρέπει να εξασφαλίσουμε. Και επίση το βασικό μήνυμα από όλε τι εκθέσει είναι για να έχουμε βιωσιμότητα χρειαζόμαστε φιλόδοξου στόχους σε ό,τι αφορά την κλιματική αλλαγή και το περιβάλλον. Δηλαδή είναι απολύτω απαραίτητο για να επιτευχθούν οι στόχοι τη βιώσιμη ανάπτυξη των ΗΠΑ στο 2030. Εφόσον βέβαια πάντοτε είμαστε σε θέση να διατηρήσουμε τη θέρμανση του πλανήτη στον 1,5 βαθμό και εφόσον είμαστε σε θέση να μειώσουμε αντίστοιχα και τι εκπομπέ μα. Και νομίζω πω η Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ είναι πρωτεργάτη. Ορίζει δηλαδή τα απαραίτητα πρότυπα σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση και Ε, καταφέρει να το κάνει ακριβώς επειδή δεν έχει και αυτά τα χαρακτηριστικά, αν θέλετε, ε, του εθνικού, αν θέλετε, εγωισμού των επιμέρους κρατώμενων. Επίσης, τώρα αναφέρθηκαν κάποιες κριτικές σε ό,τι αφορά την ε, Διακυβερνητική Επιτροπή IPCC. Εγώ όμως μπορώ να σας αναφερθώ στην οπτική γωνία με βάση την οποία αποτελεί την, τον πιο σημαντικό και αξιόπιστο μηχανισμό διήθησης, αν θέλετε, επιστημονικών δεδομένων που οδηγούν σε μια επιστημονική συνένεση, δηλαδή σε ένα επίπεδο συνένεσης μέσω του οποίου οι επιστήμονες για ορισμένα επιστημονικά πορίσματα μπορούν να μιλούν με την ίδια φωνή και να έχουν την ίδια άποψη. Και κατά τελευταία ε, εβδομάδα των διαπραγματεύσεων ε, που έγιναν ε, σε επίπεδο Ολομέλειας IPCC, στην οποία συμμετέχουν 195 κυβερνήσεις, και στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων που έλαβαν χώρα εκεί, ε, θα πρέπει να πούμε ότι πραγματικά στο πλαίσιο αυτή τη έκθεση εξετάζονται όλε οι παράγραφοι. Κάθε λέξη ουσιαστικά τίθεται υπό αξιολόγηση. Και έτσι το προϊόν τελικά που προκύπτει αποτελεί ένα κοινό αποτέλεσμα, μια κοινή προσπάθεια δηλαδή από τον επιστημονικό χώρο και τον πολιτικό χώρο. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο έχουμε ένα νέο προϊόν το οποίο δεν αμφισβητείται σε ό,τι αφορά σε επιμέρους φράσεις, σε ό,τι αφορά τις επιμέρους λέξεις. Τώρα, το κατά πόσο εφαρμόζεται στην πράξη ε, το περιεχόμενο αυτής της έκθεσης και κατά πόσο ακολουθούν τους, τις, τις, τις δεσμεύσεις τους οι κυβερνήσεις είναι ένα άλλο θέμα, γιατί πράγματι δεν βλέπουμε να, τις, να τα αποκρίνονται στις δεσμεύσεις τους. Τώρα, το κατά πόσο η ζημία για την, για την αλληλεία, αν είμαστε σε θέρμανση της τάξης των 2 βαθμών Κελσίου, αυτό θα εξαρτηθεί από την ε, κάθε περιοχή. Δηλαδή σε κάποιες ε, περιοχές ε, θα υπάρξει μείωση γιατί μία αλληλεία εξειδικευμένη σε ένα συγκεκριμένο είδος θα εξαφανιστεί ακριβώς επειδή θα έχει εξαφανιστεί το συγκεκριμένο είδος από εκείνη την περιοχή και θα μετακινηθεί αλλού. Αλλά όπως σας είπα, εάν έχουμε υψηλότερη αύξηση από τον 1,5 βαθμό, αρχίζουμε και κινούμαστε σε τελείως διαφορετικό, σε διαφορετική διάσταση. Οπότε, σε ό,τι αφορά το, την αξιολόγηση ε, του πώς θα εξελιχθούν έτσι τα οικοσυστήματα, θα πρέπει να έχουμε υποχρεωτικά πια κάποιε ζώνες στις οποίε δεν θα υπάρχει κανένα είδος αλλίευση, ώστε να γνωρίζουμε τι ακριβώς, ποιε ακριβώς δηλαδή είναι εξελίξει με βάση αμυγό και μόνο το κλίμα και τα συγκεκριμένα ε, είδη. Ερώτηση από τον πρόεδρο. Μήπως μπορείτε να αναφερθείτε και στι ε, στις ε, αν θέλετε άνθρακα, δηλαδή στα σημεία που συλλέγουν άνθρακα, carbon sinks. Μπορείτε λίγο να μας εξηγήσετε. Δέσμευση άνθρακα, έτσι. Μιλάμε για αυτές τις δεξαμενές, τα sinks. Τι είναι ακριβώς. Δηλαδή, αποθήκευση άνθρακα κάτω από τη θάλασσα. Απάντηση. Εγώ σας, ε, μπορώ να σας μιλήσω για λύσεις που βασίζονται στη φύση, όχι τεχνολογία δηλαδή το τι μπορεί να γίνει σε ό,τι αφορά τις δυνατότητες αποθήκευσης άνθρακα. Η δέσμευση λοιπόν και αποθήκευση άνθρακα για το Carbon Capture and Storage είναι, εφαρμόζεται ήδη, δηλαδή υπάρχουν ε, από τα αποθέματα φυσικού αερίου τέτοιες δυνατότητε, όπου δηλαδή συλλέγεται, συλλέγονται και αποθηκεύονται. Αλλά σε ό,τι αφορά αυτά τα σημεία και αυτή την εφαρμογή, δηλαδή συλλογή και δέσμευση και αυτέ τι σχετικέ τεχνολογίε, όσο πιο κοντά βρισκόμαστε σε ανθρώπινου οικισμού, τόσο πιο δύσκολο είναι αυτό το ζήτημα. Ναι, ήθελα να ξέρω από τεχνικής απόψεως πώς αντιμετωπίζετε αυτό. Μιλήσατε για ένα πηγάδι, μια δυνατότητα αποθήκευσης. Είναι κάτι που θα πρέπει να το συζητήσουμε και νομίζω ότι πρέπει να προχωρήσουμε. Είναι οι γεωλογικές λύσεις, κάτι που υπάρχει κάτω από τους ωκεανούς μία παρατήρηση. Είπατε στην αρχή ότι αυτό που είπα δεν είναι η προσωπική μου άποψη. Ναι, έχετε δίκιο, δεν είναι η προσωπική μου άποψη. Ήθελα όμως να σας δώσω την αφορμή να μιλήσετε για την Διακυβερνητική Επιτροπή και γιατί αυτά που λέτε είναι πολύ σημαντικά. Έχετε δίκιο. Ε, ζητώ συγγνώμη, λέει ο Πρόεδρος, πρέπει να επιταχύνουμε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, λέει η κυρία Μάτο και ευχαριστούμε και για την ε, Επιστημονική Επιτροπή για αυτήν την ε, πολύ σημαντική ε, έκθεση. Βεβαίως όλοι γνωρίζουμε ότι η, αλλαγή, η κλιματική αλλαγή, η όξυνση των ωκεανών ε, οπωσδήποτε οδηγεί σε μείωση των αποθεμάτων. Θα, θα ήταν κανείς πολύ κοντόθωρος εάν ε, όμως εστρέφω το μονάχα όσον αφορά την αποκατάσταση ε, αυτής της κατάστασης αν υπεδείκνει λέω μονάχα τους αλληλείς. Ε, νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι ότι θα πρέπει η προσέγγιση να είναι ολοκληρωμένη και υποστηριζόμενη και από την επιστήμη αλλά και από τις τοπικές κοινωνίες οι οποίες θα πρέπει να προστατευτούν βάσει αυτής της συμφωνίας ε, ε, για τις παράκτιες κοινότητες αλλά θα πρέπει να υποστηριχθεί και το Κοινοβούλιο στην εντολή που έχει όσον αφορά την πολιτική συμμετοχή. Δηλαδή δεν θα πρέπει όποιο, είτε ε, με άλλου, ε, ε, είτε με ταμεία πόρους ευρωπαϊκούς, είτε μέσα από οποιοδήποτε ταμείο συνεχής και άλλο, να υποστηρίξει τις καύσιμες, τα, καύσιμα, τα ορυκτά καύσιμα θα ήθελα να μάθω εάν έχετε κάποια στοιχεία όσον αφορά την επίπτωση που έχουν στα θαλάσσια οικοσυστήματα. Και ε, οι εξορίξεις ε, καθώς επίσης ε, και οι εξορίξεις στη θάλασσα και οι ε, Θα ήθελα να μου πείτε επίσης με ποιο τρόπο μπορεί ε, να ε, έχει επίπτωση η διαφορετική, αυτό που αναφέρατε όσον αφορά τη δικτύωση των προστατευμένων περιοχών σε σχέση και με την προστασία συγκεκριμένων ειδών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε λέει η κυρία Σαμπό. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι η έκθεση αυτή, καθώς επίσης και η έκθεση του IPBES ε, όσον αφορά ε, την κλιματική αλλαγή, έρχεται μια στιγμή που το Κοινοβούλιο θα πρέπει να πάρει απόφαση όσον αφορά την ε, χρήση ε, των ε, πόρων για υποστήριξη της αλίας, αλλά επίσης θα πρέπει να αποφανθεί και επί των αλλιευτικών συμφωνιών που η Ευρωπαϊκή Ένωση υπογράφει με τρίτες χώρες. Σε αυτά που λέτε κατανοώ δύο σημαντικά κατά την άποψή μου πράγματα. Πρώτον, ότι, ε, η, ότι η πόρη και η αλία γενικότερα επηρεάζεται ιδιαίτερα από την κλιματική αλλαγή, αλλά καταλαβαίνω ότι υπογραμμίζεται και το γεγονός ότι η ίδια η αλληλεία μπορεί να ε, αποτελέσει μέσω των απαντήσεων που μπορούν να δοθούν ε, στις κλιματικές προκλήσεις. Από τη μία πλευρά, μέσα από την ε, κάλλιστη δυνατή διαχείριση των αποθεμάτων, αλλά και ενδεχομένως μειώνοντας τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου μέσω των εκπομπών των αλλιευτικών ε, πλοίων. ...25 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα ε, διαθέτουμε ε, και επομένως εδώ οδηγούμε σε τρεις ερωτήσεις. Οι πολιτικές μας βασίζονται στα επιστημονικά στοιχεία. Ακούγοντάς σας καταλαβαίνουμε ότι τα επιστημονικά στοιχεία ε, δεν είναι βεβαία, δηλαδή ε, περιλαμβάνει ακόμα πολλά ερωτηματικά. Ε, η, ικανότητα των οικοσυστημάτων και των αλλιευτικών πόρων σχετίζονται με τη δικιά μας ικανότητα να απαντήσουμε στις κλιματικές προκλήσεις. Άρα θα πρέπει το monitoring, η επιτήρηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στα οικοσυστήματα θα πρέπει να είναι καλύτερη έτσι ώστε να επιτηρήσουμε με τη σειρά μας καλύτερα τα δεδομένα που έχουμε στις ποσοστώσεις και στα μέγιστα υποτρεπόμενα λιεύματά μας. Δεύτερον, προστατευμένες ε, περιοχές, MPAs, ε, υπάρχουν πολλές τέτοιες παράκτιες ε, περιοχές τις οποίες επιθυμείτε και που μου φαίνεται ότι μπορεί να είναι ένα πολύ καλό εργαλείο όπως είναι τα πάρκα αλλά και οι μεγάλες ευρείες προστατευόμενες περιοχές στα ανοιχτά. Τρίτον, ε, εσείς θα μπορούσατε να υποστηρίξετε ε, την υδατοκαλλιέργεια με την προϋπόθεση της βιωσιμότητας βεβαίως. Mr. Gonzalez Ο κύριος Γκονζάλης Κασάρης, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε ε, καθηγητά, για αυτή την ε, έκθεση η οποία πραγματικά μας ε, ε, υπενθυμίζει ότι συμβαίνουν ε, σημαντικές αλλαγές και επομένως θα πρέπει να πάρουμε μέτρα αποφασιστικά. Είμαι και εγώ μέλος της Επιτροπής ΕΝΒΗ, σας άκουσα και σε αυτήν την Κοινοβουλευτική Επιτροπή και οπωσδήποτε υπάρχει μεγάλη συσχέτιση ανάμεσα στα λιευτικά αποθέματα και την κλιματική αλλαγή. πρόσφατα εγκρίναμε προσχέδιο έκθεσης ε, για την COP25 όπου δεσμευόμαστε να ε, μειώσουμε κατά 55% μέχρι το 2030 τις ε, εκπομπές μας και μέχρι το 50% να έχουμε οδετερότητα εκπομπών. Μιλώντας για αλληλεία δεν είναι δυνατόν να αποφύγουμε κάποιες ερωτήσεις. Πρώτον, έχουμε παράκτιες κοινότητες οι οποίες ζουν από την αλληλεία και όπου οπωσδήποτε οποιαδήποτε αλλαγή θα τις επηρεάσει ιδιαίτερα. Ε, μια και έρχομαι από τη σοσιαλιστική ομάδα, πιστεύω ότι θα πρέπει να σκεφτούμε και αυτούς τους ψαράδες ε, και να βρούμε δίκαιους τρόπους να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα αυτά. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να λύσουμε τα προβλήματα τα οποία απορρέουν από την κλιματική αλλαγή. Συμφωνώ με τον κύριο Μιγιαμόν ότι τελικά ε, δεν είναι αίτιο η αλία, αλλά είναι θύμα βιώσιμη αλληλεία, βιωσιμότητα της αλληλείας. Αυτό προσπαθούμε ε, και επιδιώκουμε μέσα από την κοινή αλιευτική ε, πολιτική ε, που θα υποστηρίξει βεβαίως και τους ωκεανούς και τους αλιευτικούς μας τόλους. Θα ήθελα να υποβάλω και άλλες ερωτήσεις. Θεωρώ ότι το θέμα των, των προστατευομένων περιοχών είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά να υποβάλω λοιπόν τις ερωτήσεις. Θεωρείτε ότι ε, η βιοτεχνική αλληλεία θα μπορούσε να προκαλέσει προβλήματα σε σχέση και με την κλιματική αλλαγή. Και... Ε, Πιστεύετε ότι εάν υποστηριχθεί η μείωση των εκπομπών των αλλιευτικών σκαφών μέσα από την βελτίωση των κινητήρων τους ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό ε, θα μειωθούν, ε, με αυτό θα μειωθούν οι εκπομπές και επομένως θα μειωθούν και οι επιπτώσεις ε, της κλιματικής αλλαγής και κάτι άλλο. Δεν διάβασα όλη την έκθεση. Τις ερωτήσεις μπορείτε να προχωρήσετε στις ερωτήσεις. Μία ακόμα ερώτηση, αν είναι δυνατόν. Σχετικά με την κρυόσφαιρα. Ε, και οι μόνιμοι παγετώνες, αλλά και τα ε, λιγότερα χιόνια ε, στις, στα βουνά, τα οποία θα έχουν σαν αποτέλεσμα λιγότερα νερά, τα οποία σε όλη τη διάρκεια του έτους θα φτάνουν μέχρι τα δέλτα των ποταμών. Πιστεύετε ότι μπορεί να προκαλέσουν επιπλέον προβλήματα. Ευχαριστούμε πολύ. Λέει η κυρία Κέλλερ, για τα όσα μας είπατε, πραγματικά μας ε, προκαλούν ε, μεγάλο προβληματισμό όλα αυτά. Πιστεύω πάντως ότι στο Κοινοβούλιο έχουμε την ε, δυνατότητα να αναλάβουμε δράση και θα έχουμε ευκαιρίες. Πολλές ερωτήσεις έχουν ήδη υποβληθεί, είχα και εγώ μία. Όσον αφορά αυτό το θέμα της όξυνσης, της αύξησης της οξύτητας, εν πάση περιπτώσει, ε, και την μείωση του οξυγόνου. Ε, ε, ναι, μπορεί να υπάρχει αποχρωματισμός, το αναφέρατε εσείς προηγουμένως, αλλά ε, μήπως υπάρχουν και επιπτώσεις και για άλλου είδους ε, οργανισμούς. Επίσης, έχετε κάποια ιδέα σχετικά με το ποσοστό της βιοπικιλότητας ε, που θα έχει ε, πρόβλημα λόγω της αλλαγής των επιπέδων του πεχά Ωραία, αυτή ήταν πολύ συγκεκριμένη ερώτηση. Ο κύριος Γκερέρα. Ευχαριστώ. Να εκφράσω και εγώ και σχόλια. υπάρχουν κάποιες, ε, κάποια συμπεράσματα σε σχέση με τα οποία υπάρχουν διαφορετικές τοποθετήσεις σε ό,τι αφορά ε, διαφορετικές πολιτικές ομάδες. Εμείς πάντως ε, από την πλευρά της δικής μου χώρας της Πορτογαλίας δηλαδή έχουμε επηρεαστεί στις παράκτες περιοχές πολύ από την κλιματική αλλαγή και οι δικέ μα κυβερνήσει δεν έχουν λάβει υπόψη του τα επιστημονικά δεδομένα και αυτή τη συγκεκριμένα την έκθεση τη Κυβερνητική Επιτροπή. Θα ήθελα να θέσω κάποια γρήγορα ερωτήματα. Ε, στη διαφάνεια που μας δείξατε υπάρχουν κάποιες ιδιαίτερες ε, περιοχές ε, οι οποίες βρίσκονται στα κόκκινα, αλλά δεν μας έχετε αναφέρει περαιτέρω δεδομένα. Ποιες άλλες ακριβώς είναι απαραίτητες ούτως ώστε να αποφύγουμε με καλές σημείες. Μετά, σε ό,τι αφορά τα διαφορετικά σενάρια που μα αναφέρατε, σε ό,τι αφορά δηλαδή περισσότερη εξήνηση και ούτω καθεξή, σε ό,τι αφορά τι παράκτητες περιοχέ, υπάρχει μια γενικότερη άποψη, για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά για παράδειγμα την κατασκευή για παράδειγμα αερολιμένων σε παράκτητες περιοχές ε, για παράδειγμα ε, όπως έχει γίνει στην Πορτογαλία πρόσφατα ε, κοντά στις εκολές ενός ποταμού που θα μπορούσε να έχει επιπτώσεις. Γενικότερα δηλαδή η κατασκευή μηχανικών περιοχών σε παράκτητες περιοχές θα μπορούσε να έχει αυξημένες αρνητικές συνέπειες. Μετά, σε σχέση με αυτά τα σενάρια νομίζω πως θα πρέπει να υπάρξει μια πολιτική η οποία θα θέσει ε, τη σωστή προτεραιότητα και η Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να εξασφαλίσουμε για παράδειγμα την ασφάλεια της ε, διατροφικής αλυσίδας. Από εκεί και μετά ένα ακόμα, ένα ακόμα ερώτημα είναι το κατά πόσο ε, κατά πόσο υπάρχουν περαιτέρω επιπτώσεις ή ε, αυξημένες επιπτώσεις σε ό,τι αφορά ε, ύδατα σε πιο μεγάλο βάθος. Ε, κατά πόσο δηλαδή υπάρχει μια τέτοια εξειδικευμένη εμπειρογνωμοσύνη και επίση ε, ε, ποιε θα είναι απαραίτητε επενδύσει που θα πρέπει να κάνουμε ώστε ακριβώ στι ε, περιοχέ να μπορέσουμε να διατηρήσουμε τι συγκεκριμένε κοινότητε. Πρόεδρο, κύριε καθηγητά, σα δίνω το λόγο. Σας, θα σα παρακαλέσω να είστε όσο το δυνατόν πιο σύντομο γίνεται. Ναι, μπορώ να είμαι πολύ σύντομο λέει ο ε, γιατί υπάρχουν ε, κάποιες από αυτές τις ερωτήσεις ε, για τις οποίες δεν μπορώ να είμαι συγκεκριμένος και να δώσω απαντήσεις, γιατί υπήρξε μία ομάδα εργασίας, δύο της IPCC και μία ομάδα ένα. Η δύο αναφέρθηκε στις φυσικές αλλαγές, ενώ η ένα αναφέρθηκε στον ευάλωτο χαρακτήρα και στις δυνατότητες προσαρμογής των ανθρώπων. Οπότε εμείς δεν αναφερθήκαμε στις τεχνολογικές λύσεις, αλλά Αντιθέτω, η ομάδα 3 θα είναι εκείνη η οποία θα ασχοληθεί με αυτό το ζήτημα. Σε ό,τι αφορά τι δυνατέ λύσει, εμεί εξετάσαμε ποιε προσαρμογέ είναι δυνατέ σε ό,τι αφορά την ε, περιοχή των παράκτιων περιοχών, για παράδειγμα, εμ, ασύσταση των εμ, παράκτιων οικοσυστημάτων ή ε, τα αποθέματα άνθρακα και ούτω καθεξής. Εκείνο που μπορώ να σας πω είναι ότι όλοι οι κλάδοι θα πρέπει να συμβάλλουν ε, στην ε, επίτευξη των στόχων ε, των εκπομπών, δηλαδή και η αλληλεία και για παράδειγμα θα πρέπει να υπάρχει ε, υπάρξει και ουδέτερο σε ό,τι αφορά τι εκπομπέ άνθρακα στόλο. Γιατί αν θέλουμε να επιτύχουμε αυτού του στόχου στο 2030, τότε θα πρέπει να ξεκινήσουμε άμεσα. Μέσα στον επόμενο χρόνο, μέσα στην επόμενο μήνα θα πρέπει να ξεκινήσει η προσπάθεια. Αυτό δηλαδή είναι το ε, γενικό σφαιρικό μήνυμα το οποίο προκύπτει από όλες τις εκθέσει και εκείνη για τον 1,5 βαθμό και εκείνη που αφορά τις ελσέ περιοχές και εκείνη που αφορά ε, τους ωκεανού. Το βασικότερο, το σημαντικότερο μήνυμα είναι πάντοτε η μείωση των εκπομπών άνθρακα. Και αυτό μπορώ να σας πω εγώ για τη δική μας ε, έκθεση είναι ότι έχουμε κάποια κεφάλαια σε ό,τι αφορά επιμέρους περιοχές σε ό,τι αφορά αυτή την έκθεση δηλαδή της ομάδας 2 και ε, αναφερόμαστε στο, σε ένα επίπεδο ανάλυσης το οποίο δεν είναι τόσο, ε, πιο, τόσο λεπτομερές. Ε, δηλαδή, ε, στο μέλλον θα υπάρξουν κεφαλαία τα οποία θα είναι εξειδικευμένα σε ό,τι αφορά περιοχές και τους ωκεανούς συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά τις επιμέρους περιοχές. Θα υπάρχει δηλαδή στοχευμένη, εξειδικευμένη ε, πληροφορήση σε ό,τι αφορά συγκεκριμένε περιοχέ και του ωκεανού για αυτέ τι περιοχέ, ε, ειδικότερα για την Ευρώπη, όπου έχουμε τόσο μεγάλη ποικιλομορφία σε ό,τι αφορά τις παρακτές περιοχές. Σε ό,τι αφορά την επίπτωση τη ε, της οξύνησης ε, των ωκεανών, έχουμε πολύ συγκεκριμένες επιπτώσεις όπω για παράδειγμα η αποτιτάνωση, αλλά από εκεί και μετά υπάρχουν και πολύ συγκεκριμένε επιπτώσει σε ό,τι αφορά την, ε, τη θαλάσσια ζωή. Δηλαδή δεν έχουμε μόνο περίπτωση αποτιτάνωση, είναι και πιο εκτεταμένε οι, ε, οι επιπτώσει. Και αν κάνουμε μια προσωμείωση ε, εργαστηριακά στο πώς θα έχουν τα πράγματα ε, στα τέλη του αιώνα, δεν μπορούμε να προβλέψουμε το πώς θα εξελιχθεί το ένα οικοσύστημα και δεν ξέρω αν πότε θα είμαστε σε θέση να το κάνουμε, γιατί ε, σίγουρα θα είναι διαφορετική εξέλιξη αυτού του οικοσυστήματος ανάλογα με τα επίπεδα της ε, οξύνησης ε, του ωκεανού. Αλλά όπως σας είπα υπάρχουν και συνέργειες ανετικές μεταξύ θέρμανσης του πλανήτη, θέρμανσης των ωκεανών και ε, οξύνησης των ωκεανών. Αλλά και πάλι δεν μπορεί κανείς εύκολα να προβλέψει την εξέλιξη των οικοσυστημάτων. Σε κάθε περίπτωση όμω θα είναι φτωχότερα αυτά τα οικοσυστήματα, δηλαδή θα υπάρχει σίγουρα χαμηλότερη βιοπικιλότητα. Πρόεδρο. Και σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα ερωτήματα, ουσιαστικά αυτό που μα λέτε είναι ότι δεν έχετε κάποιε απαντήσει, τουλάχιστον προ το παρόν. Ναι, ε, Πρόεδρε, αναφέρθηκαν κάποια πολιτικά σχόλια σε συνδυασμό με ερωτήματα. Ε, οπότε είναι δύσκολο κανεί να διακρίνει ποιο είναι ακριβώ το ερώτημα. Αλλά εάν έχω αφήσει κάτι σε κρεμότητα, μπορώ να επανέλθω. Ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρος, ε, κύριε καθηγητά, την παρουσία σα ε, εδώ και για την παρουσίαση που μα κάνατε. Μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο σημείο λοιπόν της ημερήσιας διάταξη, ε, δηλαδή τα όρια αλευμάτων σε ό,τι αφορά τα αποθέματα στη Βαλτική. Κύριε Κώστα, που έχει επανέλθει εδώ. Δηλαδή είναι σημαντικό να παρακολουθούμε το τι συμβαίνει σε αυτέ τι συνεδριάσει όπου αποφασίζονται τα συνολικά επιτροπόμενα μετά τα τάξη. Γνωρίζουμε πω η τελευταία συνάντηση έλαβε χώρα την ε, τελευταίο μήνα προκειμένου να καθοριστούν τα τάξη αυτά για ε, τη Βαλτική. Υπήρχε, υπάρχει και ένα έγγραφο το οποίο έχει διανεμηθεί σε όλου, το οποίο περιλαμβάνει τι συστάσει του ΆΕΣΥ σε ό,τι αφορά τα τάξη που θα πρέπει να οριστούν, τι προτάσει τη Επιτροπή και το τι συμφωνήθηκε τελικά. Επίση, ζητήσαμε από τη Φιλανδική Προεδρία να παρευρεθεί σήμερα εδώ, αλλά αρνήθηκε να το κάνει η Φιλανδική Προεδρία και δεν είναι κάτι το καινούριο. Και παρότι το Συμβούλιο συχνά μας αναφέρει ότι αυτό το ζήτημα, δηλαδή τα τάξη ό,τι αφορά τη Βαλτική αποτελεί ζήτημα εθνικής αρμοδιότητας, από την άλλη πλευρά έχουμε ένα πολιετές σχέδιο αλεύσεις σε ό,τι αφορά ακριβώ την Βαλτική. Ε, και από εκεί και μετά υπάρχει και μια σχετική έκθεση από την η οποία ελπίζω πω θα έχουμε τη δυνατότητα να συντηθεί εδώ. Η κυρία Κίρχνερ λοιπόν έχει το λόγο από την Επιτροπή για να μα πει ποια ήταν τα αποτελέσματα αυτής της διαπραγμάτευσης σε ό,τι αφορά τα τάξε, τα όρια δηλαδή, αλεύσεις ε, στον, ε, στην Βαλτική. Υπήρξαν κάποια λοιπόν αποθέματα για κάποια είδη δηλαδή τα οποία ε, μειώθηκαν πολύ σημαντικά κατά 20%. Ε, συνολικά δεν έχουμε μεγάλη μείωση, αλλά υπήρξαν κάποια είδη στα οποία πραγματικά η περικοπή ήταν πολύ μεγάλη, έφτασε και στο 60%. Παρακαλώ, κύριε να έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, που μα προσκαλέσατε σήμερα εδώ για να σα ε, αναφέρουμε λίγο την απόφαση που έλαβε το Συμβούλιο σε ό,τι αφορά ε, τα συνολικά επιτρεπόμενα λίμματα στη Βαλτική για το 2020 και όπω μπορείτε να δείτε από την πολύ ε, ωραία εδώ συνολική επισκόπηση που διαβίβασε ε, η Γραμματεία ουσιαστικά το Συμβούλιο ε, έμεινε κοντά στην αρχική πρόταση της Επιτροπής και μόνο σε τρεις περιπτώσεις ε, παρεξέκλεινε από τις ε, αρχικές προτάσεις της Επιτροπής. Κα, λίγες ποσοστιαίες μονάδες. Οπότε έχουμε παραμείνει κοντά στο αρχικό MSY, δηλαδή την μέγιστη ε, βιομάζα, σε 6 από 8 συνολικά είδη και για τα δύο στα οποία δεν το καταφέραμε, ε, ήταν περιπτώσεις εκείνες όπου το ISIS πρότεινε να απαγορευτεί εντελώς η αλία. Και όπως σας είχα αναφέρει πέρυσι, όταν το ISIS προτείνει πλήρη απαγόρευση της αλίευσης και η Επιτροπή εφαρμόζει ένα πολυετές ε, ε, σχέδιο διαχείρισης και συγκεκριμένους κανόνες αλίευσης στο πλαίσιο αυτού του πολυετούς σχεδίου, παρότι μπορεί να υπάρχει κάποιο απόθεμα το οποίο επιτρέπεται να αλλιεύεται, ε, δεν ε, το θεωρούμε ως κάτι το οποίο γίνεται. Γιατί ε, ενώ έχουμε προβλέψει πολύ σημαντική μείωση της αλλιεύσης, υπάρχουν κάποια συνοδευτικά μέτρα. Δηλαδή υπάρχουν κάποιο, για παράδειγμα κάποια, κάποιες επιχειρησιακές, ε, ε, εποχικές συγγνώμη, απαγορεύσεις της σε ό,τι αφορά για παράδειγμα τον ανατολικό γάδο, τον δυτικό γάδο και σε ό,τι αφορά την δυτική Ρέγκα. Οπότε, κατά τη δική μας άποψη, το Συμβούλιο έλαβε με αυτά τα τάξη μια αρκετά υπεύθυνη απόφαση και κατέστη δυνατό να λάβει αυτή την απόφαση επειδή η Επιτροπή θα παράσχει κάποια υποστήριξη σε εκείνους οι οποίοι θα έχουν πληγεί ιδιαίτερα από τις πολύ σημαντικές περικοπές που έχουν γίνει σε κάποια είδη. Και μπορώ να σας δώσω περαιτέρω διευκρινήσεις βέβαια σε ό,τι αφορά ακριβώς αυτά τα υποστηρικτικά μέτρα που θα ε, παράσχει η Επιτροπή, αλλά θα σταματήσω εδώ και είμαι στη διάθεση των ε, μελών εδώ για περαιτέρω ερωτήσεις. Πρόεδρος. Ε, μας είπατε ότι θα υπάρξουμε στα περισσότερα από θέματα όπου θα φτάσουμε ε, στο επιθυμητό MSY μέχρι το 2020, δηλαδή τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση, αλλά ε, σε ό,τι αφορά για παράδειγμα τον Ανατολικό Γάδο, η πρόβλεψη είναι ότι δεν πρόκειται να ανακάμψει μέσα στο εκείς μέλλον, έτσι. Δηλαδή, αν κανείς δει το σύνολο εδώ της εικόνας, διαπιστώνει ότι υπάρχουν κάποια είδη τα οποία καταφέρουν να επιβιώσουν σε ό,τι αφορά την, την, την, μειωμένη διαθεσιμότητα οξυγόνου στο νερό και ούτω καθεξής, αλλά κάποια άλλα όχι. Οπότε η γενική σας εντύπωση σε ό,τι αφορά τα αποθέματα αιχθείων ε, μέσα στην Βαλτική, σε ό,τι αφορά τα επόμενα χρόνια, ποια είναι. Απάντηση από την κυρία Κίρσνερ. Ναι. Ουσιαστικά ε, με την κατάρρευση των αποθεμάτων ε, του γάδου της Ανατολική ε, Βαλτική, ε, Πραγματικά βρισκόμαστε σε μια δύσκολη κατάσταση, όχι μόνο λόγω των περιβαλλοντικών παραγόντων, οι οποίοι ασκούν πίεση σε αυτό το απόθεμα, αλλά και λόγω τη αλλείας. Και σε ό,τι αφορά ακριβώ τον Ανατολικό εδώ κάτω, ενημερωθήκαμε ότι περισσότερα είναι τα ψάρια τα οποία πλέον ε, ουσιαστικά εξαφανίζονται, δηλαδή πεθαίνουν λόγω των περιβαλλοντικών παραγόντων από εκείνα τα οποία αλλιεύονται. Και γι' αυτόν ακριβώ το λόγο η ποσόσταση που έχουμε προβλέψει ε, για τον γάδο, τα αλλιεύματα δεν θα είναι ικανά ούτως ώστε να οδηγήσουν σε μια ανάκαμψη το απόθεμα αυτού του ανατολικού γάδου. Λοιπόν, τα κράτη-μέλη είναι εκείνα τα οποία θα πρέπει να ενεργοποιηθούν και να εφαρμόσουν τις διάφορες οδηγίες ε, ε, για τις οποίες έχουν δεσμευτεί να προβούν σε κάποια ανάληψη δράση σε ό,τι αφορά δηλαδή την ποιότητα των ε, θαλασσών, ε, τα εντρικά και ούτω καθεξής. Δηλαδή παρότι έχουμε φτάσει ε, σε μια συμφωνία δεν εφαρμόζεται ακόμα από τα κράτη-μέλη. Για παράδειγμα, η περιεκτικότητα συνετρικό τη Βαλτική είναι πολύ υψηλή και υπάρχει λοιπόν ανάγκη ανάληψη δράση από τα κράτη-μέλη με βάση τα όσα έχουν συμφωνήσει τους ώστε να μειωθεί η συγκέντρωση συνετρικού στην Βαλτική και προκειμένου να μπορέσει να ανακάμψει και ο ε, Κύριε Πρόεδρε, ο κύριος Νίκολας Χέρψ ε, της δικής μου ομάδας από τη Γερμανία δεν, ήταν, δεν μπορούσε να είναι εδώ, γι' αυτό μου ζήτησε να πω κάτι εκπροσωπώντας τον λέει κύριος Μιγιανμόν το Συμβούλιο έλαβε ε, τε μέτρα άνευ προηγουμένου όσον αφορά ε, τον, ε, ανατολικό, τον βακαλάο της Ανατολικής Βαλτικής καθώς επίσης και για την Ρέγγα. Αυτό έχει βεβαίως και αλλιευτικές επιπτώσεις αλλά ε, και κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις στη Βαλτική. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει πρώτον ε, οπωσδήποτε να αντιμετωπίσουμε την ε, περιβαλλοντική πίεση με δημιουργία οικοσυστημάτων στη Βαλτική κλπ. Απ' την άλλη πλευρά όμως θα πρέπει να μειωθεί και η αλλιευτική ικανότητα με ταυτόχρονη διαχείριση των κοινωνικονομικών επιπτώσεων. Ο κύριος Χέρμπς λοιπόν τελειώνει λέγοντας ότι θα πρέπει όσο γίνεται πιο γρήγορα ε, να έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις ε, καθώς επίσης και συγκεκριμένη χρηματοδότηση από το Ταμείο ε, της Αλίας έτσι ώστε ο στόλος ο οποίος θα έχει επίπτωση από όλη αυτή την κατάσταση και θα έχει ζημιωθεί να βοηθηθεί. Ε, η πάυση είτε ε, περιοδική είτε μόνιμη ε, θα πρέπει να αφορά και τις δύο περιοχές της Βαλτικής και οπωσδήποτε τα μέτρα θα πρέπει να εφαρμοστούν και στην Δυτική και την Ανατολική Βαλτική και τα μέτρα να ληφθούν όσο γίνεται πιο γρήγορα. Αυτά ήθελε να πει ο κύριος Χέρπς τα οποία είπα εξ ονόματός του. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Σάλιβαν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μια ερώτηση προς το Συμβούλιο και την Κομισιόν. Το Συμβούλιο, το Αλληλευτικό Συμβούλιο ακολούθησε την συμβουλή τους ε, για ε, ποσόστοση ε, παρελιευμάτων 2.000 τόνων παρά για την Βαλτική παρά την αντίθετη γνωμοδότηση για μηδενικό τονάζ. Οι, φυσικές, οι αλλιευτικές ε, ικανότητες όμως υπολογίζονται βάσει και των παραλιευμάτων. Η Κομισιόν μπορεί να εξηγήσει ποια ε, επιπίας επιστημονικής και εμπειρικής βάσεως ε, έχει καθορίσει για το 2020 αυτό το τάκ παραλιεύματος όσον αφορά τον γάδο της Ανατολικής Βαλτικής. Thank ε, Η κυρία Κύρχε, να απαντήσω πρώτα απ' όλα στις ερωτήσεις. Στη δήλωση που έγινε ε, εξ ονόματος του κυρίου Χέρμπστ Χαιρόμαστε που σήμερα έχουμε τη δυνατότητα να είμαστε εδώ, αφού ε, το θέμα ήδη και η πρόταση έχει ήδη ε, υποβληθεί. Η ερώτηση, το, το, ε, το, τα μέτρα δηλαδή τα οποία είχε ζητήσει ο κύριος είναι γεγονός ότι έχει υπάρξει μια τροπολογία στο πολιετές σχέδιο διαχείρισης της Βαλτικής και εκεί γίνεται αναφορά στο Ταμείο Αλίας. Μπορούμε βεβαίως μετά να μπούμε και σε λεπτομέρειες όσον αφορά τη δεύτερη ερώτηση σχετικά ε, με το ΤΑΚ ε, ε, παραλιεύματος ποια είναι τα εμπειρικά στοιχεία ή τα επιστημονικά επί του οποίου βασίστηκε η πρόταση αυτή. Να σας εξηγήσω. Η κατάσταση και στη Βαλτική αλλά και σε άλλες θαλάσσιες ε, λεκάνες είναι ότι τα αλλιεύματα δεν είναι καθαρά. Δηλαδή ε, βάζουν τα δίχτυα τους ε, οι αλλιείς αλλά δεν πιάνουν μονάχα το σκοπούμενο αλλά και άλλα αλλιεύματα. Το ίδιο συμβαίνει και στην Ανατολική Βαλτική. Όταν λοιπόν οι αλληλείς βγαίνουν να ψαρέψουν το ευρωπαϊκό, την ευρωπαϊκή χωματίδα τότε ψαρεύουν ε, ας πούμε ή ε, αλείς που ψαρεύουν ε, σολομό ακόμα και για πελαγικά είδη οπωσδήποτε θα πιάσουν στα δίχτυα τους και κάποια άλλα λιεύματα. Θεωρούμε, εάν είχαμε ακολουθήσει την επιστολή της ISIS και είχαμε βάλει αυτό το ποσοστό να είναι μηδενικό, τότε θα είχαμε ε, προκαλέσει προβλήματα όχι μονάχα ε, στην Ανατολική ε, Μεσόγειο, συγγνώμη, Βαλτική, αλλά θα είχαμε δημιουργήσει προβλήματα και στην αλία του Καλκανίου. Στην ουσία, δηλαδή, αλλιεύουν πολλές εκατοντάδες σκάφη και ο περιορισμός τους αφορά τον Ανατολικό Γάδο εμείς ήρθαμε σε επαφή με την ISIS, ήρθαμε σε επαφή με τους ε, εμπειρογνώμονες, τους επιστήμονες και αυτοί μας είπαν ε, ποιο είναι το επίπεδο του, ε, της αναπο, του αναπόφευκτου παραλιεύματος και μάλιστα ε, οι ίδιοι ξανα... ήρθαν σε επαφή μαζί μας ε, και περιμένουμε βέβαια στις επόμενες ε, δέκα μέρες περί τα μέσα Νοεμβρίου να μας δώσουν την τελική τους γνωμοδότηση. Πάντως εμείς επί τη βάση των δικών τους προτάσεων κάναμε τους υπολογισμούς μας. Να υπολογίσουμε δηλαδή το ποσοστό που εμείς πιστεύουμε ότι μπορεί να αποτελεί το απαραίτητο, το αναπόφευκτο ε, και ανώφελο παραλίευμα. Ε, και όλα αυτά βέβαια μπορούν μόνο με υπολογισμούς ε, να υπολογιστούν. Όσον αφορά αυτά τα unavoidable by catches, έχοντας όλα τα στοιχεία, θα υποβάλουμε ε, τα ε, θέματα στο Συμβούλιο και βεβαίως το Συμβούλιο επί τη βάση των νέων στοιχείων όσον αφορά ε, τα αναπόφευκτα παραλιεύματα θα πρέπει να πάρει μια σχετική απόφαση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. to the uh, measure... Νομίζω ότι αναφερόμενοι στα μέτρα αυτά τα οποία θα συζητήσουμε συνειδητοποιώ ότι υπάρχουν πολιτικές δυσκολίες για το θέμα της ελίας του γάδου στη Βαλτική. Το θέμα είναι ότι ποιες είναι οι υποσυστώσεις, τι γίνεται στην πράξη, έτσι και αλλιώ έχουν περιοριστεί οι δραστηριότητες εκεί. Η Επιτροπή όμως παρόλα αυτά είχε πάρει την απόφαση να μειωθεί η χρηματοδότηση έτσι δεν είναι. Δεν πρόκειται για θέμα που επιβλήθηκε στην Επιτροπή λόγω προηγούμενου. Αν θέλετε, μπορώ να κάνω την παρουσίαση όσον αφορά την τροποποίηση και με αυτόν τον τρόπο θα απαντήσω και στην ερώτησή σας. Η Επιτροπή τέλος Οκτωβρίου έκανε μια πρόταση όσον αφορά αυτό το σχέδιο για τη Βαλτική με δύο τμήματα. Πριν παρουσιάσω το περιεχόμενο αυτής της πρότασης, θα ήθελα καταρχήν να σας πω ότι η Επιτροπή έχει, δίνει μεγάλη σημασία σε αυτήν την έκθεση, σε αυτή την πρόταση. Είναι κάτι πάρα πολύ επίγον, αν θέλετε. Οι αλλοί σήμερα αντιμετωπίζουν στην περιοχή της Βαλτικής μία, αν θέλετε, κατάσταση όπου έχει ε, αρχίσει να ισχύει το πλέγμα των έκτακτων μέτρων όσον αφορά την αλία του γάδου στη Βαλτική. Και βεβαίως ε, το θέμα είναι εδώ πώς θα αντιμετωπιστούν τα δύο επόμενα χρόνια, το άμεσο μέλλον δηλαδή. Είναι σημαντικό για μας επίσης να υποβάλουμε μία πρόταση η οποία να παρουσιάζει ένα διαρθρωτικό πλάνο για όλους αυτούς τους αλίες που εξαρτώνται από την αλία του γάδου στην περιοχή αυτή. Και αυτό βεβαίως θα πρέπει να προχωρήσει με ταχύτητα τους ρυθμούς στον τριμερή διάλογο. Αυτή είναι η πρότασή μας. Θα παρουσιάσω καταρχήν το κομμάτι της αλίας και ο Βενσό, ο συνάδελφος που είναι δίπλα μου, θα παρουσιάσει το κομμάτι του πολιετούς ε, χρηματοδοτικού πλαισίου. Όσον αφορά τώρα το κομμάτι της Ελίας, τι προτείναμε ακριβώς ε, σαν σχέδιο για την Βαλτική και την Ελία του Γάδου. Θέλουμε καταρχήν να συνειδητοποιήσουν όλοι ότι υπάρχει μία κατάσταση επίγουσα, γι' αυτό και υποβάλλουμε αυτά τα πάρα πολύ ε, ακριβή και αστηρά μέτρα. Όσον αφορά καταρχήν τα αλληλευτικά σκάφη, τα οποία δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Ανατολικής Βαλτικής. Τα μέτρα λοιπόν όσον αφορά τον παρεδεσιακό εξοπλισμό που χρησιμοποιούν αυτά τα σκάφη, ανώτατα όρια, τα κράτη-μέλη μέχρι τώρα χρησιμοποιούν τη χρηματοδότηση αυτή για την ε, εξάλληψη κάποιων από τα αλεαυτικά σκάφη και τα ανώτατα όρια έχουν μειωθεί πολύ σημαντικά, καθώς και ανώτατες ποσότητες για όλα τα κράτη-μέλη που δραστηριοποιούνται στην περιοχή αυτή της Ανατολικής ε, Βαλτικής. Επίσης, έγιναν πιο αυστηρά τα μέτρα και οι κανονισμοί στο τωρινό σχέδιο για τη Βαλτική έχουμε ποσότητες οι οποίες ε, εκφορτώνονται σε πολύ συγκεκριμένες τοποθεσίες. Δεν μπορεί κάποιος να εκφορτώσει όπου θέλει, ε, όποια και να είναι, αν θέλετε, η επιθυμία του. Υπάρχουν συγκεκριμένα σημεία εκφόρτωσης με συγκεκριμένους τρόπους παρακολούθησης, εποπτείας και ελέγχου των εκφορτώσεων. 50 κιλά από τη στιγμή δηλαδή που κάποιος έχει 250 ε, ε, κιλά αλλιεύματος μπορεί και πρέπει είναι κάτι το οποίο σαφώς ε, και θα καθοριστεί βάσει των νέων μέτρων τις περιοχές, 6 ναυτικά μίλια, 25 με 30 είναι ο, μίλια είναι ο καθορισμός των περιοχών και βεβαίως προκαθορίζονται και οι εξοπλισμοί και ο τρόπος ελέγχου και επιτήρησης με ηλεκτρονικό τρόπο. Υπάρχει εδώ η συγκεκριμένη κατανομή των ποσοτήτων, η παρατήρηση. Βεβαίως δεν γίνεται έλεγχος σε κάθε συγκεκριμένο σκάφος. Περίπου 25% των σκαφών ελέγχονται. Αυτά όσον αφορά την αλληλεία. Θα δώσω τώρα το λόγο στον συνάδελφο, ο οποίος θα μιλήσει για το θέμα της χρηματοδότησης. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε και κύριοι. Όπως εξήγησε η συνάδελφος Μάγια, υπάρχει μια τροπολογία όσον αφορά το πολιετές πρόγραμμα διαχείρισης ε, της ε, ε, Βαλτικής που αφορά ε, και το, το, το γενικότερο πλαίσιο 14-19. Στόχος είναι η, η στα πλαίσια του άρθρου 34 του εν λόγω κανονισμού να εισαχθεί μέτρο ε, οικονομικής υποστήριξης ε, που θα αφορά την τελειωτική πάυση. Ε, είχε εκπνεύσει η προηγούμενη διορία. Το μέτρο αυτό αφορά αποκλειστικά τα λιευτικά σκάφη τα οποία ιδιαίτερως εξαρτώνται από την ελεία του γάδου της Ανατολικής Βαλτικής. Οι προϋποθέσεις ε, είναι αυτές οι οποίες προβλέπονται ε, εις ε, το άρθρο 34 του κανονισμού ΕΤΘΑ. Αφορά την μακροπρόθεσμη εξισορρόπηση της αλίευσης σε σχέση με, την διαθέσιμη, με τους διαθέσιμους αλιευτικούς πόρους. Εδώ προστίθεται και μια τροπολογία η οποία δίνει την δυνατότητα να αναμοφλευχθούν τα ε, ποσά τα οποία είχαν δοθεί αρχικά στην ε, αποθήκευση και την διαχείριση των ε, πόρων έτσι ώστε να δίνεται η δυνατότητα από το 2014 μέχρι το 2019 να χρησιμοποιηθούν οι πόροι αυτοί για τους λόγους τους οποίους ανέφερα προηγουμένως. Ευχαριστώ πολύ. Thank you. wish to speak? Εγώ σας ευχαριστώ. Θέλει κάποιος να πάρει το λόγο. Όχι από ό,τι φαίνεται. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόταση. Βεβαίως ε, θα προσπαθήσουμε να προχωρήσουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα, έτσι ώστε να διευκολύνουμε και εμείς την πρόοδο, αλλά καταλαβαίνετε ότι εδώ ε, μιλάμε ε, για σημαντικά πράγματα. Μιλάμε βέβαια και για κάτι το οποίο θα συζητηθεί ενδεχομένως το Δεκέμβριο και επομένως θα ψηφιστεί ίσως τον Φεβρουάριο, τον Μάρτιο στην Ολομέλεια. Θα το δούμε. Θα πάντως σας βεβαιώ ότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε έτσι ώστε να προχωρήσει το θέμα όσο γίνεται πιο γρήγορα. Πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ ε, πάρα πολύ κυρία Κνίσνερ ε, ε, και θα σας ε, περιμένουμε ξανά ε, το, τον Φεβρουάριο, το Δεκέμβριο, συγγνώμη, έτσι ώστε να μας πείτε ε, ποια, ποιες θα είναι οι προτάσεις σας για την μέγιστη επιτρεπόμενη απόδοση για το 2020. Γιατί πώς είναι δυνατόν να συνεδριάσει η Επιτροπή μας χωρίς εσάς. Περνάμε στο επόμενο θέμα, παρουσίαση ε, ε, των εργασιών της Επιτροπής Ελέγχου ε, των Αλλιευμάτων. Έχουμε εδώ τον Πρόεδρο, κύριο Πασκάλ Σαβουρέ. Νομίζω ότι όλοι γνωρίζετε ποιο είναι το έργο αυτής της υπηρεσίας και θα σας δώσω το λόγο κύριε Σαβουρέ. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ που μας καλέσατε σήμερα για να παρουσιάσουμε τις υπηρεσίες μας στο έργο. Έχω παρουσιάσει για την περίοδο 2024 ένα πρόγραμμα εργασιών το οποίο θα παρουσιάσω καθώς και τις επιδόσεις για το 2019, ένα έτος το οποίο δεν έχει ολοκληρωθεί. Θα συνεχίσω στα γαλλικά. Όπως ξέρετε, πρόκειται για μια υπηρεσία, την υπηρεσία ελέγχου της Αλίας, που δημιουργήθηκε το 2005 μετά από απόφαση του Συμβουλίου με την πρόταση υπαριθμών 2005 κάθετος 3261 πρόκειται για μια αποκεντρωμένη υπηρεσία η οποία κωδικοποιήθηκε το 2019 473 με σκοπό την επιτήρηση των δραστηριοτήτων αλίας και την συνεργασία στον τομέα της αλίας για να τηρούνται οι κανονισμοί και η υλοποίηση των κοινών πρακτικών αλίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα σας παρουσιάσω σήμερα την δράση της υπηρεσίας μας. Θέλω όμως να σας ε, υπενθυμίσω ότι το γνωστό ως Joint Deployment Plan, κοινό σχέδιο ανάπτυξης, συντονισμός ε, ουσιαστικά των δραστηριοτήτων ε, των ε, κρατών μελών με σκοπό την καλύτερη επίτευξη των δραστηριοτήτων ελέγχου. Θέλω να σας πενθυμίσω ότι το 2018 κάναμε 27.000 ελέγχους, 3.000 στη θάλασσα και 650 παράτυπες δραστηριότητες εντοπίστηκαν πολλές φορές εξαιρετικά σοβαρές. Η δραστηριότητά μας για τον έλεγχο κάθε παράτυπης και μη ελεγχόμενης δραστηριότητας αλίας, καθώς και η προσπάθεια στήριξης ε, βάσει των προγραμμάτων ελέγχου και επιτήρησης σε συνεργασία με τις άλλες διευθύνσεις και υπηρεσίες, η στήριξη επίσης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνεωριοφυλακής και Ακτοφυλακής της Frontex αλλά και της, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα και για να μιλήσουμε λίγο και για τα μέσα που διαθέτουμε από την Ευρωπαϊκή Αρχή προϋπολογισμού διαθέτουμε για το 20 17,6 εκατομμύρια ευρώ, 0,7 στα πλαίσια του προγράμματος PESCAO που το οποίο σας ανέφερα προηγουμένως. Είμαστε 60 άτομα. Θα προσλάβουμε αρχές Ιανουαρίου του 20 και ένα καινούριο συνεργάτη. 44% γυναίκες. Θα επανέλθω σε αυτό σε λίγο, διότι αναφέρεται εξάλλου και στην έκθεση απαλλαγή τη υπηρεσία μα το θέμα αυτό τη εκπροσώπησης των δύο φύλων. Έχουμε ένα διοικητικό συμβούλιο με ένα εκπρόσωπο ανακράτος μέλος και έξι εκπροσώπους Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επίσης έχουμε και ένα συμβουλευτικό όργανο, συμβουλευτικό ε, συμβούλιο, βάσει της ε, κοινής πολιτικής της Αλίας Σκοπός αυτού του συμβουλευτικού οργάνου είναι η στήριξη του εκτελεστικού διευθυντή όσον αφορά την διεκπαιρέωση των ελέγχων, της επιτήρησης, αλλά και η συνεργασία με τους μη κυβερνητικού οργανισμούς. Για να επικεντρωθώ λίγο στα μέσα που διαθέτουμε, το 2018 η εκτέλεση του προηγουμένου έφτασε το 98,7% το ποσό της εκτέλεσης των πληρωμών 87,6% και θα ήθελα εδώ να προσθέσω ότι πραγματικά εκτελέσαμε τον προϋπολογισμό μας κατά 98%. Όσον αφορά το ελεγκτικό συνέδριο για τα στοιχεία του 2018 είχαμε μία έκθεση χωρίς παρατηρήσεις, κάτι που είναι πολύ θετικό. Κάθε πέντε χρόνια υπάρχει η περιοδική αξιολόγηση των επιδόσεων της ε, υπηρεσίας και βεβαίως ε, οι συστάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου υλοποιούνται ε, αμέσως μετά την περιοδική αξιολόγηση. Η τελευταία έλαβε χώρα το 2016, η πρώτη το 2011-12. Υλοποιούμε δηλαδή ε, τις ε, συστάσεις της αξιολόγησης που έγινε το 2016-17. Είμαστε μια μικρή υπηρεσία, προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε όσα μέσα διαθέτουμε με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο και να υπογράψουμε συμφωνίες συνεργασίας με άλλες υπηρεσίες, με τη Frontex, με την EMSA, με τον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Έχουμε πάνω από 25 συμβάσεις για την παροχή υπηρεσιών με άλλους οργανισμούς και υπηρεσίες που ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πάνω από 60 συμβάσεις πλαίσιο στα πλαίσια των δραστηριοτήτων μας έχουν συναυθεί με άλλους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και όσον αφορά το προσωπικό, τις διαδικασίες, έχουμε υιοθετήσει όλα τα συστήματα της Επιτροπής, ABAC, CISPER 2, Είμαστε σε πολύ καλή, αν θέλετε, σειρά όσον αφορά την υλοποίηση αυτών των συστημάτων για την παρακολούθηση των αποστολών μας. Τώρα, 19 διαφορετικές εθνικότητες εκπροσωπούνται στην ε, υπηρεσία μας. 44% ε, είναι το ποσοστό εκπροσώπησης των γυναικών. Τα τελευταία χρόνια σε όλους τους ευρωπαϊκούς ε, οργανισμούς και θεσμούς. Έχει υποβληθεί μείωση των μέσων καθώς και περικοπές 11% όσον αφορά τη δική μας ε, υπηρεσία. Σήμερα λοιπόν διαθέτουμε 61 ε, εργαζόμενους εκ των οποίων τρεις χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα ΠΕΣΚΑΟ. Το θέμα τώρα της ίσης εκπροσώπησης ε, των δύο φύλων. Εμείς εφαρμόζουμε εδώ όλους τους κανονισμούς, ε, όπως και όλοι οι ευρωπαϊκοί θυσμοί για τις άδειες μητρότητας, γονικές άδειες, ευελιξία. Δεν προσπαθούμε δηλαδή απλώς να διευκολύνουμε την ε, εργασία των γυναικών, αλλά θέλουμε να δώσουμε και κάποιες δυνατότητες ε, ε, των ε, υπαλλήλων μας, εξάλλου απευθυνόμαστε σε όλους τους υπαλλήλους, άνδρες και γυναίκες, για να υπάρξει μία δυνατότητα ειδικών αδειών σε περίπτωση οικογενειακών υποχρεώσεων. Τα θέματα των παρενοχλήσεων στο χώρο εργασίας, θέλουμε να επιτύχουμε μια ισορροπία μεταξύ της οικογενειακής και της επαγγελματικής ζωής. Γι' αυτό και υλοποιούμε όλα τα μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση. Για τις προσλήψεις, κάθε νέα πρόσληψη γίνεται έχοντας κατά νου την ε, ίση εκπροσώπηση των δύο φύλων, έτσι ώστε να αποφύγουμε κάθε στρέβλωση και κάθε είδους διάκριση στις προσλήψεις μας. Το 2016 38% ήταν οι γυναίκες εργαζόμενες, το 2019 44%. Οι επικεφαλής τμήματων, οι υποδιευθυντές η εκπροσώπηση των γυναικών ήταν πάνω από 40% στο διοικητικό προσωπικού. Έχουμε φτάσει σχεδόν το 50%, ενώ το 2016 η εκπροσώπηση των γυναικών σε αυτές τις διευθυντικές θέσεις ήταν μόνο 20%. Ε, παρακολουθούμε λοιπόν και υλοποιούμε τις συστάσεις και προτάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εδώ βλέπετε μια φωτογραφία του προσωπικού μας. Η οργάνωση είναι πολύ απλή. Έχουμε τρία τμήματα. Μία για την πληροφορική, το προσωπικό, την ασφάλεια και το περιβάλλον. Δύο επιχειρησιακές ε, ε, μονάδες, Βόρειος Ατλαντικός και οι δραστηριότητε Κατά καταπολέμησης παράτυπης αλίας και η υλοποίηση και συνεργασία με τα προγράμματα ΠΕΣΚΑΟ και άλλα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε τον εκτελεστικό διευθυντή, το συμβουλευτικό όργανο και το διοικητικό συμβούλιο. Για το 2019 ο προπολογισμός 17,4 εκατομμύρια, 8 για το προσωπικό, διοικητικές διαπάνες πάνω από 6 εκατομμύρια, 6,9 συν η επιδότηση για το πρόγραμμα ΠΕΣΚΑΟ. Για το 2020 το σχέδιο προϋπολογισμού, κάτι που είχε την θετική άποψη του Διοικητικού Συμβουλίου, 6,9 για το προσωπικό, 6 για την πληροφορική, διοικητικά έξοδα, ενίκιο, 6,7 εκατομμύρια συνεισφορά στο πρόγραμμα Πεσκάου 680.000, σύνολο 17,5 εκατομμύρια για το 2020. Δραστηριότητες ε, επιχειρησιακές. Βλέπετε, διαβάζοντας το πρόγραμμα δραστηριοτήτων μας, ότι έχουμε τέσσερις επιχειρησιακές δραστηριότητες. Καταρχήν το JDP, το ενιαίο πρόγραμμα ανάπτυξης, ανάπτυξη κοινή βάση του προγράμματος αυτού, δεύτερον ε, αξιολόγηση κινδύνου, ανάλυση δεδομένων, τρία το πρόγραμμα Πεσκάο και κάθε είδους παρακολούθηση προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά πολέμηση της ε, παρατυπιζαλίας και άλλες διεθνείς δραστηριότητες. Όπως βλέπετε, έχουμε ένα ευρύ φάσμα γεωγραφικής κάλυψης, έξι διαφορετικά κοινά προγράμματα ανάπτυξης, τα ευρωπαϊκά Βαλτική, Βόρεια Θάλασσα, ήταν εξάλλου και το πρώτο πρόγραμμα μας το 2007, δυτικές περιοχές, Μεσόγειος, εύξηνος πόντος με δύο κρατημέλη καθώς και συνεργασία με τρίτες χώρες που ξεκίνησε πέρσι. Βόρεια Ατλαντική, ελεγχόμενες περιοχές, σε πάνω, σε πάνω στα γαλλικά. Δεν θα σας δώσω τώρα όλα τα αλλιεύματα, γιατί βλέπετε ότι έχουμε 38 διαφορετικά είδη ιχνιών σε αυτά τα, αποκαλύπτονται από αυτά τα κοινά προγράμματα ε, αλλιευμάτων όσον αφορά τον έλεγχο των ευρωπαϊκών αρχών. Σήμερα και εδώ θα ήθελα να σας αναφέρω τα συνολικά ε, αλλιευτικά σκάφη 77.500 αλλιευτικά σκάφη, ε, ε, τράτες 10.388, 13,4%, άλλου είδους 3.591, 4,6% ε, και τα υπόλοιπα είναι στατικού είδους αλλιευτικά αλλιευτικοί εξοπλισμοί. 82, μάλιστα σχεδόν 83% ε, του στόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελείται από ε, ε, σκάφη μεγαλύτερα από 12 μέτρα. Ναι, υπάρχουν όμως και σκάφη τα οποία ε, ε, ξεφεύγουν από οποιοδήποτε έλεγχο και κυρίως τους κανόνες ελέγχου που υφίστανται όλα τα σκάφη. Ε, επίσης, η υπηρεσία για να προχωρήσει σε αυτούς τους ελέγχους, εκτός από τους ίδιους πόρους, χρησιμοποιεί και 2.000 Ευρωπαίους επιθεωρητές που έχουν την δυνατότητα να κάνουν και την πιστοποίηση, να κάνουν τέτοιου είδους είδους ε, ε, επιθεωρήσεις. 3.000 δε επιθεωρήσεις έγιναν στη θάλασσα. Ε, θέλω τώρα να αναφερθώ ε, στο θέμα της συμβολής των κρατών μελών. Ε, 2.612 ημέρες περιπολία περιπολίας, 657 ώρες πτήσης και θαλάσσιας επιτήρησης καθώς επίσης ε, ε, και 200 ε, περίπου ανταλλαγές επιθεωρητών, σχεδόν δηλαδή χίλιες ημέρες επιθεώρησης όσον αφορά την τυποποίηση και την διαφάνεια μεταξύ των κρατών μελών. Θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι το 2018 το συνολικό κόστος των ελέγχων, των αποστολών ελέγχων της κοινή ανάπτυξης που έγιναν δηλαδή και από τα κράτη-μέλη καθώς επίσης και από την υπηρεσία όσον αφορά το κόστος έφτασε τα 78 εκατομμύρια ευρώ. Όπως μπορείτε να διαπιστώσετε εδώ, η τάση λόγω της αύξησης του ΑΕΠ αλλά καθώς ε, ε, και κάποια είδη πλέον επιτηρούνται από το πρόγραμμα κοινή ανάπτυξης οδηγεί στην αύξηση, την σταθερή αύξηση από το 2013 και ένθεν των ε, κοινών επιθεωρήσεων. Φτάσαμε τώρα σε 27.000 συντονισμένες ε, επιθεωρήσεις. Ε, και η τάση αυτή η αυξητική επιβεβαιώνεται. όσον αφορά τις παραβιάσεις, το 2018 παραβιάσεις ή υποψία παραβίασης ε, που θα πρέπει να επιβεβαιωθεί από τα κράτη-μέλη ε, έφτασε ε, στις 6.000 σοβαρές παραβιάσεις ενώ τώρα οι αριθμοί έχουν αυξηθεί ακόμα περισσότερο. Η τυπολογία τώρα των παραβιάσεων, όπως και πέρσι, μάλλον όπως και στο παρελθόν, στην ουσία αντιμετωπίζουμε ε, προβλήματα τα οποία σχετίζονται είτε με ελλειπή είτε με ε, πλήρη έλλειψη αναφοράς ε, αλλιευμάτων καθώς επίσης ε, και ελλειπή μέτρα ε, τεχνικής συντήρησης. Ε, άλλες παραβιάσεις αφορούν τους βρόχους, αφορούν το μέγεθος των βρόχων, την χρήση και ανάπτυξη των δικτυών, καθώς επίσης και τις υποχρεώσεις εκφόρτωσης. Επίσης, στα διεθνή ύδατα αντιμετωπίζουμε παρόμοια κατάσταση, αλλά εκεί έχουμε και προβλήματα τα οποία αφορούν την διαχείριση. 3.000 έρευνες επιθεωρήσεις ε, στη θάλασσα ε, εκεί αντιμετωπίσαμε και συγκεκριμένες περιπτώσεις ε, παρεμπόδισης και παρακόλλησης της επιτήρησης, ε, ενεργητική δηλαδή παρακόλληση και παθητική παρακόλληση επίσης. Εδώ θα ήθελα να πω ότι το JDP, το πρόγραμμα δηλαδή κοινών, το, κοινό πρόγραμμα ανάπτυξης ξεκίνησε μετά από μάλλον ε, βάσει αυτών των κοινών προγραμμάτων ε, κινητοποιούνται ποινικέ εθνικές διαδικασίες. Ε, θα, θα έπρεπε να είχα ήδη αναφέρει ότι στα πλαίσια των αποστολών συνεργασίας και συντονισμού η υπηρεσία μας επικουρεί και τις ομάδες περιφερειακού ελέγχου. Ε, είναι αυτές οι ομάδες οι οποίες επιβλέπουν την περιφερειοποίηση. Προχωρούν ε, σε διαδικασίες ε, αξιολόγησης ε, ε, κινδύνου, εφαρμογής ε, των συστημάτων και των περιορισμών της εκφόρτωσης. Επίσης έχουμε δουλέψει από κοινού στην αξιολόγηση της συμμόρφωσης, κυρίως όσον αφορά πάλι τις εκφορτώσεις. Επίσης η υπηρεσία διαχειρίστηκε ομάδα εργασίας σχετικά με τις, ε, ε, τις τεχνολογίες ηλεκτρονικής ε, τηλεεπιτήρησης. Αναφέρομαι τώρα εις τα θέματα τα οποία ξεπερνούν την, τα συστήματα επιχειρησιακής συνεργασίας ε, και να αναφερθώ συγκεκριμένα στην αξιολόγηση κινδύνου και την ανάλυση δεδομένων. Κάθε χρόνο ε, λαμβάνει ε, χιλιάδες στοιχεία VMS από τις χώρες μέλη, καθώς επίσης και στοιχεία VAS που ε, δίνουν την, ε, μας δίνουν την ε, δυνατότητα να αναλύσουμε τις δραστηριότητες αλίευσης και βάσει των στοιχείων που έχουμε και των αναλύσεων που κάνουμε προχωρούμε σε περιφερειακές βελτιώσεις έτσι ώστε η έλεγχη να είναι καλύτερα στοχευμένη και στις πιο ευαίσθητες περιοχές μάλιστα. Επίσης έχουμε συνεργαστεί με τα κράτη-μέλη έτσι ώστε να αναπτύξουμε κοινέ διαδικασίες αξιολόγησης κινδύνου έτσι ώστε ε, τα κράτη να δουλεύουν με παρόμοιο τρόπο όσον αφορά προβληματικές οι οποίες ε, ε, είναι παρόμοιες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όσον αφορά τον, το στρατηγικό πεδίο 3, την διεθνή διάσταση δηλαδή, εδώ συζητούμε περισσότερο για την συνεργασία με τα κράτη-μέλη, αλλά εδώ δουλεύουμε περισσότερο και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υποστηρίζουμε δηλαδή την Κομισιόν στην διεθνή της ε, διάσταση της κοινή ελευθερικής πολιτικής και να πω εδώ ότι καμία ε, καμία ε, κίνηση δεν μπορεί να κάνει, καμία δράση δεν μπορεί να αναπτυχθεί ε, σε, διεθνή, σε διεθνές περιβάλλον εάν δεν έχει προηγουμένως πράσινο φως από την Κομισιόν. Ε, εδώ υλοποιούμε και το άρθρο 30 υπό την αίρεση των υπολείπων νομικών στοιχείων που αναφέρει ότι οι σχέσεις με τις τρίτες χώρες οπωσδήποτε θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη και την περιφερειοποίηση έτσι ώστε να γίνονται σεβαστά, ε, ε, σεβαστές όλες οι διεθνείς συμφωνίες. Δουλεύουμε λοιπόν με την Κομισιόν, δουλεύουμε επίσης ε, και πάντα σε σεβασμό του κανονισμού για την παράνομη άναρχη κλπ. Ε, συνεργαζόμαστε με την Κομισιόν και για την καταπολέμηση της ελευθερία και παράνομης ε, αλίας σε τρίτες ε, χώρες, καθώς επίσης ε, είμαστε παρόντες στις συνεδριάσεις ε, των ε, περιφερειών Αλίας. Το πρόγραμμα είναι πενταετές, θα ολοκληρωθεί το 2022 και αποτελεί πραγματική επένδυση σχεδόν 2,6 δις, εκατομμυρίων συγγνώμη, και έχουμε δύο υποεπιτροπές ε, η υποεπιτροπή για την ε, ε, Μαυριτανία, την Σενεγάλη, τη Σιέρα Λεόν, την Γουινέα κλπ. Καθώς επίσης και μία άλλη είναι η SRFC και μετά έχουμε και την Επιτροπή αλληλία της Δυτικής Κεντρικής, του Δυτικού Κεντρικού Κόλπου της Γουινέας. FCWC. Ε, η δράση μας ευθυγραμμίζεται με τρεις άξονες. Ε, πρώτον, νομική ευθυγράμμιση ε, των ένομων τάξεων αυτών των χωρών με τις διεθνείς συνθήκες. Δεύτερον, κατάρτιση επιθεωρητών. Τρίτος άξονας, τεχνική υποστήριξη Όσον αφορά ε, την, ε, τα συστήματα παρακολούθησης ε, σκαφών, έχουμε επίσης συμβάλει σε επιθεωρήσεις και δράσεις τις οποίες έχουν οι ίδιες αυτές οι χώρες καθοδηγήσει και πρέπει να πω ότι έχουν στεφθεί από επιτυχία αυτού του είδους οι αποστολές. Θα ήθελα τώρα να φτάσω πλέον ε, στο τελευταίο πεδίο δράσεων της ε, υπηρεσίας μας, δηλαδή αυτό που αφορά την ενίσχυση των ικανοτήτων και την συνεργασία με την ακτοφυλακή. Ευρωπαϊκή ακτοφυλακή. Η ε, δράση αυτή ήταν ιδιαίτερος επωφελής και για την υπηρεσία αλλά και για την αλλιευτική κοινότητα. Ε, γιατί ε, και σε συνεργασία με την ΕΜΣΑ και με την Frontex πολλαπλασιάσαμε κατά την άποψή μου επί 20 αν όχι επί 30 το επίπεδο πληροφόρησης. Επίσης είχαμε... Et par ailleurs, nous avons pu bénéficier et nous bénéficions euh, des moyens aériens. Ε, ε, ε, χρησιμοποιήσαμε, τα, επωφεληθήκαμε μάλλον από τα ενιαία μέσα του Frontex. Ε, η Ευρωπαϊκή Ακτοφυλακή είναι μια ιδέα η οποία βασίζεται σε 11 ε, δράσεις ε, που αφορούν ε, όχι μόνο την αλληλεία αλλά και την καταπολέμηση του, της μόλυνσης, τα τελωνία, την βοήθεια προς τα πλοία, την, τις διαδικασίες διάσωσης στη θάλασσα και οι συνομοθέτες αποφάσισαν ε, να δώσουν τη μορφή του ε, κανονισμού και ε, να δώσουν την υποστήριξη μέσα από πέντε δράσεις των τριών υπηρεσιών ΕΦΚΑ, ΕΜΣΑ και Frontex που αφορούν την διοίκηση, την ακτοφυλακή κλπ. Όλους αυτούς δηλαδή που δρούν στα πλαίσια της προστασίας των θαλασσών για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε αυτές τις δεσμεύσεις και για να μπορέσουμε να δουλέψουμε με, τις, τους 316 ε, οργανισμούς, ο νομοθέτης ε, θεώρησε σκόπιμο ε, να καθορίσει πέντε πεδία εργασίας για ό,τι αφορά ας πούμε τα συστήματα επιτήρησης κυρίως δορυφορικής, την διαμήραση ικανοτήτων, για την ώρα πλοίων και αεροπλάνων, αργότερα ίσως και drones. Ε, επίσης, διαδικασίες ανάλυσης κινδύνου από κοινού, από τις ε, τρεις ε, οντότητες, έτσι ώστε να γίνεται πολυεπίπεδη ανάλυση κινδύνου, την διαμήραση πληροφοριών, και στα πλαίσια αυτού του πεδίου η υπηρεσία έχει να ναυλώσει ε, σκάφος ε, που σκοπό έχει να προχωρήσει σε ελέγχους ε, που αφορούν την αλληλεία, αλλά επίσης και να συμμετάσχει σε διαδικασίες έρευνας και διάσωσης όταν αυτό είναι απαραίτητο και χάρη στη συνεργασία με την ΕΜΣΑ την δυνατότητα μέτρων κατά της μόλυνσης. η συνεργασία τώρα με τα κράτη-μέλη. Είτε στα πλαίσια ελέγχου αλίας, είτε και στα πλαίσια της εκτοφυλακής, ο άξονας αυτός είναι πάρα πολύ σημαντικός και αποτελεί κύριο άξονα των δραστηριοτήτων μας. Ε, πρέπει να σας πω ότι ε, την ε, προηγούμενη χρονιά έχουμε καταρτήσει 600 ε, περίπου επιθεωρητές ε, από χώρες εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε προχωρήσει σε διαδικασίες διδασκαλίας εξ αποστάσεως. Έχουμε ένα σύστημα με βίντεο Επίσης έχουμε εκδώσει εγχειρίδιο το οποίο αφορά την συνεργασία με την ακτοφυλακή. Εδώ βλέπετε τη φωτογραφία ενός σκάφους, το ανέφερα προηγουμένως, όμως δεν χρειάζεται να μην πω τίποτα παραπάνω. Θα ήθελα να πω και κάτι το οποίο συχνά ξεχνούμε για να ε, υλοποιηθούν όλα αυτά τα επιχειρησιακά προγράμματα. Ε, υπάρχουν και οι άνθρωποι οι οποίοι ε, καλύπτουν τις πιο διοικητικές ας πούμε πράξεις. Έχουμε συνεργασία και επικοινωνία όσον αφορά ε, τις δράσεις μας. Δουλεύουμε με τα κοινωνικά δίκτυα. Όσον αφορά την επικοινωνία προσπαθούμε όσο είναι δυνατόν ε, να φέρουμε πιο κοντά την Ευρωπαϊκή Ένωση στους πολίτες, αλλά προσπαθούμε και να επικοινωνήσουμε ε, σε τοπικό επίπεδο και στην Ισπανία κυρίως σε περιφερειακό επίπεδο. Σε επίπεδο δηλαδή περιφερειών. Ε, ε, βεβαίως όλες οι δράσεις ε, χρειάζονται και διοικητική υποστήριξη ε, και επομένως το, τα διοικητικά συμβούλια θέλουμε να δουλεύουν με τον κάλλιστο δυνατό τρόπο. ο προπολογισμό, το οργανόγραμμα των υπαλλήλων καθορίζονται από και ελέγχονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Είναι σημαντικό η υπηρεσία επίσης να είναι παρούσα και να συνεργάζεται με άλλους οργανισμούς και υπηρεσίες. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εμείς θέλουμε να γίνουν γνωστές οι δυνατότητες και οι υπηρεσίες που μπορούμε ε, να προωθήσουμε έτσι ώστε να είμαστε χρήσιμοι στους πολίτες και τέλος ε, χρειαζόμαστε ε, δόκιμες υπηρεσίες, αποτελεσματικές υπηρεσίες έτσι ώστε να μπορέσουμε να επιτύχουμε το ικανοποιητικό ποσοστό εκτέλεσης του προπολογισμού το οποίο ανέφερα καθώς επίσης και να επιτύχουμε και τους στόχους όσον αφορά την συμμόρφωση και την δεοντολογία έτσι όπως αυτά ορίζονται από τα ε, νομοθετικά κείμενα. Ε, η ΕΦΚΑ είναι μικρή υπηρεσία, αλλά ε, είμαστε εξαιρετικά αποφασισμένοι να δουλέψουμε καλά Έχουμε καλή οργάνωση χρόνου εργασίας, ε, θέλουμε να βελτιώσουμε την συμμόρφωση μέσα από κοινά προγράμματα, προσπαθούμε να επιτύχουμε ε, καλύτερη ε, και πιο δίκαιη ίση αντιμετώπιση των εμπορευομένων και να έχουμε μια ασφαλή θαλάσσια στρατηγική. Ε, το θέμα της βιωσιμότητας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η συμμόρφωση ε, είναι ένας τρόπος να ε, επιτραπεί ή να οδεύσουμε προς τη βιωσιμότητα των πόρων. Ε, οι ικανότητές μας μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για την επιτήρηση προστατευόμενων περιοχών και τέλος όσον αφορά την διαδικασία φύλαξης ε, των ε, ακτών εμείς συμμετέχουμε στην διαδικασία της ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα τελειώσω με ένα στοιχείο το οποίο αποτελεί περισσότερο αίτημα η υπηρεσία θα ευγνωμονούσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εάν ε, μπορούσε να υποστηρίξει ε, την δυνατότητα της ε, υπηρεσίας να είναι επιλέξιμη έτσι ώστε να μπορέσει να έχει πιο αποτελεσματική οικονομική διαχείριση και περισσότερους πόρους. Ευχαριστώ πολύ. Thank you, uh, Ευχαριστώ πολύ, το Γενικό Διευθυντή. So thank you, uh, You've been in the job about years now. Um, thank you for the presentation. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ και 8 χρόνια έχετε αυτή τη θέση. Μπορείτε να μας μιλήσετε για τη συμμόρφωση, γιατί αύριο έχουμε μια ακρόαση για το θέμα αυτό των ελέγχων και θα πάρετε το λόγο. Μπορείτε να μας πείτε ποια είναι τα κράτη-μέλη που τηρούν τους κανόνες και ποια ε, λιγότερο. Έχετε αποτελέσματα. Εννοείται όσον αφορά τον ηλεκτρονικό έλεγχο εξωποστάσεως. ποια είναι τα κράτη-μέλη που τηρούν καλύτερα τους κανόνες. Δεν μπορώ να σας απαντήσω, κύριε Πρόεδρε. Η στρατηγική, αν θέλετε, αξιολόγηση του κινδύνου δεν βασίζεται στις ε, σημαίες. Έχουμε άλλες παραμέτρους. Τα συγκεκριμένα στοιχεία βασίζονται, αν θέλετε, στις ποσότητες, στα αλλιεύματα, στον εποχιακό χαρακτήρα αυτών των στοιχείων και όχι στην σημαία του σκάφους. Αναφερόμαστε σε άλλου είδους κατανομή των στοιχείων. Και όλη αυτή, αν θέλετε, η προσέγγιση μας, αξιολόγηση του κινδύνου βασίζεται σε αυτό. Πώς μπορούμε όμως να πιέσουμε τα κράτη-μέλη να τηρήσουν τους κανόνες και η Επιτροπή μπορεί να εντοπίσει ε, πώς τηρούνται οι κανόνες όταν, παραδείγματο χάρη, καλείται να αναθεωρήσει την νομοθεσία, τη, τους κανονισμούς. Αυτή η ερώτηση, αν θέλετε, βασίζεται στο γεγονός ότι τα κράτη-μέλη είναι αυτά που πρέπει να ανατρέξουν ε, στις ε, ε, σημαίες των σκαφών και στο κατά πόσο υπάρχει δεν υπάρχει συμμόρφωση. Αυτό δεν είναι δουλειά της υπηρεσίας. Θα έπρεπε όμως. Κονσάλες Κασάρες, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Γενικέ Διευθυντά. Πριν από λίγες εβδομάδες είχα την δυνατότητα, την ευκαιρία να επισκεφθώ την έδρα της ε, υπηρεσίας και από πρώτο χέρι να δω τις δραστηριότητες. Η εκτίμησή μου είναι ότι δεν, μπορεί να γίνει, δεν μπορούν να γίνουν πολλά με λίγα. Ε, είναι, ε, εδώ μιλάμε για την υπηρεσία ε, η οποία έχει το χαμηλότερο προπολογισμό και κάθε τόσο, κάθε χρόνο διευρύνονται οι αρμοδιότητές της. Με αυτή την ε, προπολογιστική, τέλο πάντων δημοσιονομική πίεση δεν είναι δυνατόν. Η ΕΦΚΑ πάντως παίζει σημαντικό κεντρικό ρόλο στην αρχιτεκτονική της αλληλείας λόγω του ελέγχου, της επιτήρησης, της επαγρύπνησης ε, η επαγρύπνηση, η πίεση που ασκεί είναι πάρα πολύ σημαντική για την κοινή αλληλευτική πολιτική και για τη διατήρηση των αλληλευτικών πόρων. Επίσης ε, είναι ουσιαστική και για την ε, ε, εκπλήρωση των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης. Οπωσδήποτε πολλά ακόμα πρέπει να γίνουν. Βεβαίως δεν, πρόκειται να δεν είναι δυνατόν να προστίθενται συνέχεια στόχοι αλλά είχαμε θετική εξέλιξη τα τελευταία χρόνια, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να έχουμε τα πλήρη αποτελέσματα βάσει του, των νέων κανόνων για τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση για το 2020 και, εν πάση περιπτώσει, όταν θα μπορέσει και η υπηρεσία να φτάσει ε, στο μέγιστο επίπεδο ε, επιτήρησης και ελέγχων, τότε θα έχουμε οπωσδήποτε καλύτερα αποτελέσματα. Ε, θα είναι γεγονός ότι θα πρέπει ο προγραμματισμός να είναι πολυετής και ότι θα πρέπει ε, να δοθούν ε, και βοήθειες όσον αφορά ε, τους πόρους. Τέλος, θα ήθελα να πω στον Πρόεδρο, τον κύριο Ντέιβις, ότι θα μπορούσαμε να εκπλαγούμε βλέποντας ότι οι χώρες οι οποίες περισσότερο συμβάλλουν είναι αυτές οι οποίες αλλιεύουν περισσότερο και αυτέ δίνουν και τα περισσότερα στοιχεία. Κύριε Πρόεδρε, σα ευχαριστώ πολύ κύριε Διευθυντά για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Έχω μια πάρα πολύ απλή και συγκεκριμένη ερώτηση επιπλέον αυτών που ήδη ακούστηκαν. Υπάρχουν περιοχές, ή ζώνες αλίας ε, στην Ευρώπη που είναι πολύ πιο δύσκολο να επιτευχθεί έλεγχος ή αλλού που είναι πιο εύκολο και πώς μπορούμε να εναρμονίσουμε τη συνεργασία και τις διαδικασίες με τις τοπικές αρχές. Στην έκθεση που μας παρουσιάσατε αναφερθήκατε στο θέμα των ε, εκφορτώσεων και των υποχρεώσεων που ρυθμίζουν αυτές τις εκφορτώσεις, αυτό αποτελεί για σας επιπλέον φόρτο εργασίας. Πρόκειται για μια δραστηριότητα, ο έλεγχος των εκφορτώσεων που γίνεται με ικανοποιητικό τρόπο στην Ευρώπη σήμερα. Είστε ικανοποιημένοι. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον κύριο Κασάρης για την ε, ερώτησή του. Όσον αφορά τη δεύτερη ερώτηση, ναι, υπάρχουν κάποια λιμάνια στην Ευρώπη που κατά κάποιο τρόπο αντιδρούν ε, έντονα στους ελέγχους, σε κάθε είδους ελέγχους. Και αυτό είναι, αν θέλετε, πιο πολύ ε, θέμα κοινωνικής ευαισθησίας και όχι τόσο πολύ συμπεριφοράς κάποιων μεμονωμένων αλλιών στη θάλασσα. Ε, δεν είχαμε πάντως γενική αντίθεση στους ελέγχους που κάνουμε κάπου ε, σε κάποιο συγκεκριμένο μέρος στην Ευρώπη. Αύριο θα επανέλθω αφού με καλέσατε στην ακρόαση που οργανώνεται. Θα επανέλθω λοιπόν στο θέμα αυτό. Και θα σας πω ότι το θέμα των απορρίψεων και την απαγόρευση για τις απορρίψεις. Εδώ πρόκειται για κάποια συγκεκριμένα αλλιεύματα, ιδιαίτερα όταν ε, πρόκειται για πάρα πολύ μικρά, ε, μικρούς ε, ηχθείες. Όμως, ο έλεγχος σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να γίνει, αν θέλετε, 24 24 ώρο και η παρακολούθηση δεν μπορεί να γίνεται από τη στιγμή που θα υπάρξει η δραστηριότητα της ΛΕΣ μέχρι τη στιγμή της απόρριψης. Και σε κάθε περίπτωση αναφερόμαστε εδώ όχι σε έλεγχο, αλλά σε μία δυνατότητα παρακολούθησης, κάτι που επαναλαμβάνω δεν μπορούμε να το διεκπαιρεώσουμε 24 ώρες, 24 ώρες σε όλες ε, τις ε, δραστηριότητες αλίας. Είναι, καταλαβαίνετε, αδύνατον με τα μέσα που διαθέτουμε. Γι' αυτό και η υπηρεσία υποστηρίζει την προσέγγιση ότι θα πρέπει να επικεντρωθούμε στις πιο ε, επικίνδυνες, θα έλεγα, περιοχές, έτσι ώστε τα συστήματα παρακολούθησης εξ αποστάσεως, όχι μόνο με ε, την ε, ύπαρξη κάμερας, αλλά και με συστήματα και την ύπαρξη και τοποθέτηση αισθητήρων. Νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο θα είμαστε πολύ πιο αποτελεσματικοί ε, στους ελέγχους μας. Θα επανέλθετε αύριο. Ευχαριστώ πολύ, ο Πρόεδρος. Έχετε ερώτηση? Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ένα, δύο μάλλον σύντομα ερωτήματα θέλω να θέσω. Καταρχήν, σε ό,τι αφορά ε, την συμμόρφωση διαφορετικών κρατών μελών με τις ε, διατάξεις. Ε, προφανώς αντιλαμβάνομαι ότι θέλετε να δεν επιθυμείτε εσείς τώρα, δείξτε με το δάχτυλο συγκεκριμένα κράτη-μέλη τα οποία ίσως να μην συμμορφώνονται σε μεγάλο βαθμό, αλλά ίσως θα μπορούσαμε να το θέσουμε αλλιώ. Θεωρείτε πως υπάρχουν διαφορές σε ό,τι αφορά τη συμμόρφωση με τους κανόνες ανάμεσα στα διαφορετικά κράτη-μέλη. Δεύτερο ερώτημα. Ποιο είναι το σημαντικό ή σημαντικότερο αίτιο για τη μη συμμόρφωση από την πλευρά των κρατών μελών με από τι διατάξει. Έλλειψη ικανοτήτων, χαμηλέ επενδύσει από την πλευρά των κρατών μελών στι ε, υπηρεσίε και τι υποδομέ ελέγχου τι είναι εκείνο που φταίει. Και κάτι τελευταίο, Πρόεδρε. Συνέχεια αναφερόμαστε στην ε, μείωση του γραφειοκρατικού άχθους ε, και την απλούστευση της νομοθεσίας. Το refit προφανώς αποτέλεσε ένα πάρα πολύ σημαντικό στόχο και ακριβώς σκόπευε στο να μειώσει την γραφειοκρατικοποίηση για τις επιχειρήσεις. Εδώ όμως στον τομέα της αλληλείας, αυτό που μας λένε οι αλληλείς είναι ότι αντί να υπάρχει λιγότερη γραφειοκρατία για ε, είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται όλο και με περισσότερη γραφειοκρατία. Άρα λοιπόν εσεί που είστε αρμόδιο από την πλευρά δηλαδή τη υπηρεσία ελέγχου τη Ένωση για την Αλία, τι θεωρείτε πώ θα πρέπει να κάνουμε ούτως ώστε να διευκολύνουμε λίγο τη ζωή των Αλία. Πώ μπορούμε δηλαδή να μειώσουμε αυτό το γραφειοκρατικό άχθο ε, και όλη αυτή την πληθώρα διατάξεων με τις οποίες ε, καλούνται να συμμορφωθούν. Σας ευχαριστώ πολύ για την ερώτησή σας. Η Κομισιόνα έχει προτείνει αναθεώρηση του κανονισμού ελέγχου και πιστεύω ότι αυτό ε, που οπωσδήποτε είναι μια διαδικασία που τους επόμενους ε, μήνες και σε σχέση με το χρονοδιάγραμμά σας, σε συνάρτηση με το χρονοδιάγραμμά σας θα υποβληθεί και στο Κοινοβούλιο, είναι ένα βήμα ε, σημαντικό όσον αφορά τη διαδικασία απλούστευσης. Επίσης, ε, ε, οι συνομοθέτες ε, ενέκριναν και υιοθέτησαν πρόσφατα κανονισμό για τα τεχνικά μέτρα, όπου ζητούν από τα κράτη-μέλη να πάρουν τεχνικά μέτρα σε περίπτωση που κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο. Με την εξέλιξη του κανονισμού ελέγχου και με τον νέο κανονισμό που μόλις ανέφερα, ε, διαμορφώνεται πλέον ένα νομικό απλουστευμένο περιβάλλον ή εν πάση περιπτώσει που οδεύει προς την απλούστευση. Δεύτερον, όσον αφορά τις συμπεριφορές και τις παραβιάσεις. Η δήλωση, η απο συγγνώμη, η έλλειψη, η απουσία δήλωσης ή η ε, ελλειπής εσφαλμένη δήλωση ε, ε, μπορεί όντως να σημαίνει ότι έχει αλλιεύσει κάποιος μεγαλύτερες ποσότητες. Άρα στο ημερολόγιο καταστρώματος προφανώς δεν θα έχει καταγράψει τα ακριβή ποσά. Πρόκειται για ένα πρόβλημα ε, το οποίο είναι πολύ σημαντικό καθότι εξαρτάται το εισόδημα του αλλιέα από το αλλιευμά του. Θα πρέπει να πιστεί ο κλάδος ότι προς το συμφέρον του είναι να αλλιεύει σύμφωνα με τους κανόνες, γιατί όταν το κάνει αυτό ε, σέβεται και τις αρχές διαχείρισης, καθώς επίσης σέβεται και την ε, δυνατότητα βιωσιμότητας όχι μονάχα του ίδιου του αλλιευτικού πόρου, αλλά και της δικής του οικονομικής βιωσιμότητας. Αναφέρθηκα προηγουμένως και σε τεχνικά μέτρα. Πιστεύουμε ότι αυτός ο νέος κανονισμός για τα τεχνικά μέτρα θα επιφέρει τροποποίηση της συμπεριφοράς, ε, καθότι θα πρέπει όλοι ε, μετά από κάποια μεταβατική διορθώνω, θα πρέπει όλοι να συμμορφωθούν με αυτά τα νέα μέτρα. Αυτή η, η μετάβαση, αυτή η τροποποίηση είναι απαραίτητη. Thank you. inaccurate declarations of catches. Ε, ε, αυτό το φαινόμενο των ανακριβών ε, αναφορών των αλευμάτων αλλιευμάτων είναι συχνό φαινόμενο ή όχι. Ναι, γιατί δεν είναι ακριβής, είτε δεν είναι ακριβής γιατί δεν έχουν ε, σωστά στοιχεία όσον αφορά το είδος ε, του αλλιεύματος ή γιατί υπάρχει υπεραλία. Το θέμα είναι λοιπόν αν υπάρχει λόγος να μην δηλώσει κανείς την ακριβή ποσότητα ε, αυτού του αλλιεύματος είτε αν το να δηλώσει λανθασμένα στοιχεία, διαφορετικά δηλαδή είδη, του επιτρέπει να αυξήσει τις ποσότητες. Η κοινή αλλιευτική πολιτική έχει πάρα πολύ ε, συγκεκριμένους στόχους όπως τη βιωσιμότητα της Το θέμα είναι λοιπόν αν ο τομέας τηρεί αυτές τις ε, κατευθυντήριες γραμμές, αυτούς τους στόχους και δηλώνει πραγματικά ε, τα αλλιεύματα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να υπάρξουν ε, ηλεκτρονικά, ηλεκτρονικά συστήματα καταγραφής ναι, αυτά τα ε, τα ηλεκτρονικά logbooks, τα ηλεκτρονικά ημερολόγια καταστρώματος. Ουσιαστικά αυτή τη στιγμή αυτό που γίνεται είναι μια δήλωση. Από τη στιγμή που υπάρχει ανθρώπινη παρέμβαση, μπορεί κάποιος να είναι ακριβής, αξιόπιστος ή λιγότερο αξιόπιστος. Γι' αυτό και οι επιθεωρήσεις, οι έλεγχοι επιτόπου, είτε την ώρα που γίνεται η εκφόρτωση, είναι πολύ σημαντική. Και εκεί συγκρίνουμε τα στοιχεία. Αυτά τα οποία ουσιαστικά έχει δηλώσει το συγκεκριμένο αλλιευτικό σκάφος σαν ποσότητες και να τα συγκρίνει με τις πραγματικές ποσότητες τη στιγμή της εκφόρτωσης. Ευχαριστώ πολύ. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσίαση αυτή, κύριε Σλάγμα. Νομίζω ότι για θέματα διαφάνειας είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρουμε ποια είναι τα στοιχεία και να μπορούμε να συγκρίνουμε τα στοιχεία των κρατών μελών. Πώς μπορούμε να κάνουμε σχόλια και παρατηρήσεις ενώ δεν ξέρουμε ποιος κάνει τι σε αυτό το τομέα. Αν κοιτάξει κανείς τα στοιχεία τα συνολικά, διαπιστώνει ότι υπάρχουν στη Βόρεια Θάλασσα πάρα πολλοί έλεγχοι και πολύ λίγες παραβιάσεις. Είναι λοιπόν αυτή η κατάσταση όπως παρουσιάζεται ακριβής. Βλέπουμε ότι υπάρχουν περιοχές με λιγότερες παραβιάσεις από άλλες. Αυτό εξαρτάται στον χαμηλό αριθμό ελέγχων. Δηλαδή, όταν κάποιος παρατηρεί πολύ λίγες παραβιάσεις σε μια περιοχή, αυτό δεν θα έπρεπε να οδηγήσει σε μείωση του αριθμού των ελέγχων. 95 παραβιάσεις βλέπω εδώ και πάνω από τριπλάσιο αριθμό ελέγχων, ενώ βλέπουμε ότι οι παραβιβάσεις μειώνονται. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν σε τι βασίζεται ε, αυτή η παρουσίαση στοιχείων. Απάντηση. Κοιτάξτε, οι παραβιάσεις, ο αριθμός των παραβιάσεων είναι ένα από τα στοιχεία, ένα σημαντικό ε, αριθμό που διαθέτουμε, γιατί οι περισσότερες από αυτές τις παραβιάσεις είναι σοβαρές. Υπάρχουν και άλλες δευτερεύουσες, θα έλεγα. Δεν μπαίνουν δηλαδή στην κατηγορία των σοβαρών παραβιάσεων. Αν κοιτάξει κανείς τον αριθμό των ελέγχων, ε, μπορώ να σας πω ότι εδώ πρόκειται για μια δειγματοληπτική ε, εικόνα που έχουμε, μια εικόνα του τομέα. Δεν θέλω να πω ότι στην Ευρώπη υπάρχει εκτεταμένη παράτυπη αλία, αλλά όταν γίνεται μια δήλωση, πολλές φορές η ακρίβεια των στοιχείων ε, δεν είναι αυτή που θα επιθυμούσαμε. Η υπηρεσία δεν έχει, αν θέλετε, στη δράση της ποινικό χαρακτήρα. Μετά εξαρτάται από την ομοθεσία των κρατών μελών το τι θα ακολουθήσει. Εμείς έχουμε ένα σύστημα αξιολόγησης βάσει κάποιας βαθμολογίας. Από εκεί και πέρα όμως, η συγκεκριμένη αντίδραση των εθνικών αρχών που μπορεί να φτάσει μέχρι και την κατάσχεση του σκάφους, εξαρτάται από τη βαρύτητα των ποινών, από την αυστηρότητα των ποινών και μετά αυτό εξαρτάται, επαναλαμβάνω, από το κάθε κράτος μέλος, από την πολιτική και την ομοθεσία ε, και το βάρος των κυρώσεων του κάθε κράτους μέλους. Ξέρετε ότι είστε εδώ χωρίς να το θέλετε, γιατί ανήκετε στο κόμμα του Brexit. Αλλά πραγματικά θέλω να σας πω ότι εγώ είμαι πάρα πολύ ευχής που σας βλέπω. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Γλυκό αυτό από μέρους σας που είπατε. Κύριε Σαβουρέ, εγώ θα ήθελα να ακούσω τη δική σας άποψη. Εσείς ως εκτελεστικός ε, διευθυντής της Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλίας ε, θεωρείτε ε, πως η επιβολή νέων ενισχύσεων του EMFF προκειμένου να δημιουργηθούν αλληλευτικοί στόλοι με σκάφη ακόμα και μεγαλύτερα από 50% είναι κάτι το οποίο έρχεται και σε αντίθεση με, τις, ε, με τους κανόνες ε, του ΟΗΕ και αποτελεί κατάχρηση, κατασπατάληση των κοντιλίων της Ένωσης. Κατά τη δική μας άποψη, με αυτή την πολιτική παραγνωρίζουμε το γεγονός ότι γενικά η αλληλευτική προσπάθεια που γίνεται ανά τον κόσμο υπερβαίνει τα αποθέματα κατά τρει έως πέντε φορές. Ε, δηλαδή, για μία ακόμα φορά ξεχνούμε τα ίδια τα ψάρια και τις μικρές κοινότητες για τις οποίες δημιουργήθηκαν αυτά τα μέτρα, δηλαδή αλληλείς οι οποίοι δεν έχουν απαραίτητους σπόρους και θέλουν να έχουν πρόσβαση σε αυτές τις αλληλευτικές ε, δυνατότητες. Ε, όλα αυτά τα καινούργια σκάφη που θα τα κάνουν όλα και θα έχουν όλες αυτές τις ικανότητες και θα αυξήσουν τις ικανότητες ε, του σκόλου που θα αλλιεύουν όταν εμείς θα έχουμε εξέλθει, ε, δηλαδή θα έχει λάβει χώρα το Brexit και από εκεί και μετά δεν θα έχετε πρόσβαση σε αυτά τα ύδατα ο πρόεδρος, ε, θέλετε να έχετε αυτά τα κονδύλια σε ό,τι αφορά τον αλληλευτικό στόλο το, ε, και τις ενισχύσει του MFFF, αλλά αυτό σημαίνει ότι τα κονδύλια δεν ε, κατευθύνονται προς τη δική σας υπηρεσία. Πηγαίνουν αλλού. Τι έχετε να πείτε, ο κ. Νομίζω πως εμείς δεν ανήκουμε σε αυτό το κομμάτι της χρηματοδότησης του του, του Υπάρχει ένα κομμάτι που αφορά την ε, Σύμβαση των Μένων Αθήνων σε ό,τι αφορά τις ε, κανόνες στη θάλασσα, που αφορά περισσότερο στον έλεγχο και ε, πρόκειται για ένα παλαιότερο κανονισμό 866 του 2006 που αργότερα ήρθε και προσθέθηκε στο Ταμείο. Και εδώ δηλαδή όταν κάνουμε λόγο για το MFF, δεν κάνω λόγο λοιπόν για την αύξηση όχι του ελευτικού στόλου, αλλά αντιθέτω, υποστήριξε από πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε ό,τι αφορά αυτό το κομμάτι, δηλαδή το επιλέξιμο σε ό,τι αφορά τι δραστηριότητε ελέγχου τη αλίας. Όχι σε ό,τι αφορά το κομμάτι του Ταμείου Θαλασσιαλίας που αφορά στο στόλο αυτό καθ' αυτό. Ε, ναι, ο κύριος Κόρμπετ ε, και άλλοι, ε, γιατί ομιλούν συνέχεια και δεν είναι ευγενική όταν εγώ παίρνω το λόγο. Εγώ όταν μιλάτε εσείς, όταν παίρνετε το λόγο, ε, σας ακούω πάντοτε και είμαι ε, ε, ε Κύριος Μιλαμών. Ευχαριστώ. Χαίρομαι πάρα πολύ που είναι εδώ ο κύριος Σαβουρέ. Και εγώ εκπροσωπώ εδώ τον ε, και την περιοχή του Βίγο, γιατί εκεί έχει την έδρα της ε, η υπηρεσία και χαίρομαι διπλά γι' αυτό. Και πραγματικά και εγώ θα ήθελα ε, να έχουμε μία υπηρεσία με περισσότερες δυνατότητες. Θυμάμαι ότι η κυρία Τομά, που η το με τους ελέγχους πάντα έλεγε ότι θα πρέπει ε, να ενισχυθούν οι έλεγχοι και να, έχουν, να διατίθενται και περισσότεροι πόροι. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν θέλω να προδικάσω τόσο θα συζητηθούν ε, αύριο, αλλά πάντως έχουμε ε, πλέον, ε, είναι σαφές ότι υπάρχει έλλειψη ομοιομορφίας. Κάθε χώρα κάνει διαφορετικά πράγματα όσον αφορά τον έλεγχο. Θα μπορούσα να πω ότι αυτόν τον χαλαρό, αυτό το χαλαρό κείμενο το ερμηνεύει ο καθένας κατά το δοκούν. Συζητήθηκε το θέμα αυτό ε, και πριν ε, από κάποιους μήνες ε, και αφιερώθηκε το 15% του προϋπολογισμού για την συλλογή και διαχείριση των επεξεργασία των δεδομένων. Ήδη στην εντολή δηλαδή αναφέρεται αυτό και δεν νομίζω ότι το Κοινοβούλιο άλλαξε αυτό το ποσοστό. Επίσης, ε, χαίρομαι γιατί αναφερθήκατε σε αυτό το ήδη διεθνές περιβάλλον, την ε, πρωτοβουλία Πεσκάο, τώρα έχουν προσθεθεί και άλλες χώρες, η Σενεγάλη, η Μαυριτανία κτλ. Αυτά είναι όλα πολύ θετικά πράγματα. Τέλος, αναφερθήκατε στο σημείο 4, στο πεδίο 4 αυτό της ε, ε, δραστηριότητας συνοριοφυλακής. Ε, με ποιους πόρους θα ολοκληρώσετε τη διαδικασία αυτή, γιατί μας είπατε προηγουμένως ότι οι πόροι είναι συγκεκριμένοι και πώς γίνεται η συνεργασία με τους άλλες δύο υπηρεσίες, δηλαδή με πώς αυτοί οι τρεις οργανισμοί συνεργάζονται. Ε, γιατί εντάξει, βλέπετε, ε, αναφέρεστε σε δραστηριότητα ακτοφυλακή, αλλά ποιοι είναι οι φυσικοί πραγματικοί πόροι τους οποίου χρησιμοποιείτε. Ε, Επίση, σε σχέση με το νέο κανονισμό έλεγχο, τα είπε προηγουμένω και ο συνάδελφο Μπελαμή, το θέμα των εκφορτώσεων, όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά, αλλά θα τα πούμε αύριο αυτά. Δεν θέλω να τα συζητήσουμε από σήμερα. Απλώ μια ερώτηση έκανα τώρα. Ε, κυρίως όσον αφορά, θέλω να μου απαντήσετε, στο θέμα με, τους, ε, ε, με την ακτοφυλακή. Ευχαριστώ πολύ. Ε, κοιτάξτε, στο, στο πεδίο 4 έχουμε προϋπολογισμό 6,2 εκατομμύρια ευρώ. Αλλά αυτός είναι ο συνολικός προϋπολογισμός που αφορά, μάλλον που περιλαμβάνει και την μισθοδοσία. Θέλω να υπογραμμίσω ότι στην ουσία ο προϋπολογισμός, από αυτό χρησιμοποιούμε 4,5 δις για να αναβλώνουμε τα σκάφη. Οπωσδήποτε είμαστε πολύ μακριά από τον μελλοντικό προϋπολογισμό του Frontex, που θα έχει 5 δις αν κατάλαβα καλά. για να δημιουργήσει την Ευρωπαϊκή Ακτοφυλακή ε, και δύο δις ε, για να υποστηρίξει τις χώρες ε, όσον αφορά τον έλεγχο εμάς, το δικό μας επίπεδο. Είναι πολύ πιο ταπεινό, ωστόσο μας ενδιαφέρει πάρα πολύ και έχουμε πραγματική βούληση να καλύψουμε αυτές, αυτά τα καθήκοντά μας. Θέλετε να απαντήσετε, κύριε Μιλιόνμον. Κοιτάξτε, εδώ είδα ε, αυτό το σκάφος ε, και είδα και αυτά που, άκουσα και αυτά που μας είπατε ε, και γι' αυτό έλεγα εάν έχετε κάποια φυσικά μέσα. Τώρα κατάλαβα ότι τα φυσικά μέσα δεν είναι δικά σας, αλλά τα αναβλώνετε, τα νοικιάζετε. Ε, τώρα όσον αφορά τη σύγκριση των ποσών που μόλις ακούσαμε, τι να σας πω, δεν, μπορούμε να, δεν μπορεί να γίνει σύν, ε, από την άλλη πλευρά, σύγκριση. Από την άλλη πλευρά η άσκηση ε, διαδικασιών λειτουργιών συνοριοφυλακής, συγγνώμη, ακτοφυλακής προφανώς δεν είναι ε, κυρίαρχο στοιχείο του, της εντολής. Από την Κομισιόν, αν έχετε να κάνετε κάποιο σχόλιο, νομίζω, παρακαλώ. Καταρχήν, θα ήθελα να συγχαρώ την υπηρεσία εδώ για την εξαιρετική δουλειά που έχει κάνει την ΕΦΚΑ και όπως ε, μόλις παρουσίασε και ο εκτελεστικός ε, διευθυντής ε, βλέπουμε πως η ΕΦΚΑ έχει υπάρξει δραστήρια σε μια σειρά από μέτρα που είναι πολύ σημαντικά σε ό,τι αφορά τη σωστή εφαρμογή της κοινής αλληλευτικής πολιτικής τόσο ε, για τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και σε ό,τι αφορά τις τρίτες χώρες, τη διεθνή δηλαδή διάσταση της αλευτικής εμπορική. Και επίσης ε, είναι πολύ σημαντικό σε ό,τι αφορά ε, τα όσα κάνει, είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος της ΕΦΚΑ σε ό,τι αφορά τις παράκτητες περιοχές. Και βέβαια εκείνο που σχετίζεται και με το επόμενο σημείο της σημερινής διάταξης που θα εξετάσουμε είναι το γεγονός ότι υπάρχουν ε, νέα και διευρυμένα καθήκοντα τα οποία ανατίθενται στην ΕΦΚΑ τα οποία θα πρέπει βέβαια να συμμορφώνονται και με το βασικό στόχο τη ΕΦΚΑ, που είναι ο συντονισμό των προσπαθειών μεταξύ των κρατών μελών σε ό,τι αφορά του ελέγχου και τι επιθεωρήσει στα ενωσιακά ύδατα. Και αυτό βέβαια αποτελεί ένα ζήτημα που θα πρέπει να μα απασχολήσει και στο ε, μέλλον και θα πρέπει να πω ότι ο κύριος ε, Πασκάλ Σαμπουρέ και η ε, ομάδα του έχουν καταφέρει να κάνουν μια μεγάλη προσπάθεια, δηλαδή και να επιτυγχάνουν περισσότερα με λιγότερα κονδύλια στη διάθεσή τους και πραγματικά είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με, την, με τις επιδόσεις της ΕΦΚΑ. Αυτά από την κοινή μας πλευρά και θα είμαστε εδώ. Ναι, ήταν πολύ καλό ο έλεγχό σα, έτσι δεν είναι κύριε Σαμπουρέ με τι σχολικέ σα επιδόσει. Κύριε Εκτελεστική Διευθυντά, εάν δεν έχετε άλλα σχόλια θα σας δούμε αύριο στο πλαίσιο της ακρόασης για τους έλεγχους. Απάντηση. Όχι, σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας, για την παρουσία μου εδώ και βέβαια αύριο θα έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε ε, και τις υποχρεώσεις εκφόρτωσης και το σχετικό σύστημα της απομακρυσμένης παρακολούθησης. Εάν θέλετε κύριε Σαβουρέ μπορείτε να παραμείνετε για το τελευταίο σημείο της σημερινής σας διαταξής για σήμερα, δηλαδή την απαλλαγή για την ΕΦΚΑ για το 2018. Ο κύριος Γκονσάλες Κασάρες λοιπόν έχει το λόγο Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Όπως ε, είπα και προηγουμένως. Νομίζω ότι πολλά δεν, δεν μπορεί να γίνονται συνέχεια περισσότερα με όλο και λιγότερα. 17 εκατομμύρια ευρώ είναι ο προϋπολογισμός ε, με ε, πιο διευρυμένες αρμοδιότητες. Έχουμε πάντως εκτέλεση περίπου 100% όσον αφορά λήψη υποχρεώσεων, 99,7% όσον αφορά δε τις υποχρεώσεις πληρωμών, 87,6%. Πρόκειται ε, για αύξηση κατά 23% των συναλλαγών πληρωμών ε, χωρίς ε, προσφυγή σε χρήση πρόσθετων πόρων, αυτό που λέγαμε προηγουμένως δηλαδή. Ε, έχουμε και καλή εκτέλεση όσον αφορά τις δραστηριότητες, 98% ε, και με ταυτόχρονη ε, αύξηση, με ταυτόχρονο συντονισμό 26.900 επιθεωρήσεων, αύξηση δηλαδή 28,46%. Το 2018 83% των πράξεων που υλοποιήθηκαν από ναυλωμένα μέσα πολλαπλού σκοπού ε, ε, αφορούσαν κυρίως την Μεσόγειο θάλασσα. Αυτό καταδεικνύει την συνέργεια με τον Frontex και με την ε, Υπηρεσία Ασφαλείας των Θαλασσών με πολύ ικανοποιητικό τρόπο. Εγώ θα υποβάλω όμως κάποιες ε, τροπολογίες, κυρίως όσον αφορά ε, την ε, καταπολέμηση της παρενόχλησης στον χώρο εργασίας, επίσης όσον αφορά τη βελτίωση της διαφάνειας ε, κυρίως δήλωση συμφερόντων του ε, εκτελεστικού διευθυντή και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου όσον αφορά την ε, σύγκρουση συμφερόντων, καθώς επίσης και την συμμόρφωση με τους κανόνες ISO 9001. Ε, ε, επίσης ε, θα προτείνουμε καταρτήσεις όσον αφορά την κατάρτιση επιθεωρητών από διάφορες χώρες. Υπάρχουν και άλλα θέματα τα οποία μπορούν να βελτιωθούν όπως ας πούμε είναι η ισόρροπη εκπροσώπηση φύλων. Θα δούμε, μας υποσχέθηκαν βελτιώσεις, διορθώσεις, γι' αυτό θα δούμε ε, και όπως λέμε και στα γαλλικιακά, μόιτας γκράσιας ε, για την εργασία σας. Any from members? Σχόλια, λέει ο Πρόεδρος. Όχι, ναι, η Κομισιόν. Θα έχετε να κάνετε σχόλια, Κομισιόν. Τα είπαμε αυτά πριν ε, από ένα μήνα περίπου όταν είχε εγγραφεί το θέμα της απαλλαγής στον προϋπολογισμό και ολοκληρώσαμε την παρέμβασή μας λέγοντας ότι η Κομισιόν είναι ιδιαίτερος ικανοποιημένη και ε, πραγματικά επενεί την ε, υπηρεσία καθότι ε, έχει για το 2018 99,7 συμμόρφωση όσον αφορά τις αναλήψεις υποχρεώσεων και 98% όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού ε, και των δραστηριοτήτων. Να υπογραμμίσω ότι ο αυξανόμενος όγκος καθηκόντων της ε, ε, υπηρεσίας σε πολλαπλούς τομείς είναι τροφή προσκέψη γιατί οπωσδήποτε θα πρέπει να ακολουθηθεί από ε, κατάλληλους ε, οικονομικούς ε, πόρους. Συμπερασματικά πάντως να πω ότι είναι πλήρης η ικανοποίηση της Κομισιόν όσον αφορά την εργασία της, της υπηρεσίας. Πάρα πολύ ωραία. Τροπολογίες μέχρι την Τετάρτη το μεσημέρι. Και με αυτό θα ολοκληρώσουμε τη σημερινή συνεδρίαση. Παρακαλώ να φέρετε αύριο ε, τι να μην λησμονήσετε να φέρετε τις ε, κάρτες σας, γιατί θα έχουμε ψηφοφορία. 9.45 θα ξεκινήσει, 9 όμως θα ξεκινήσουν οι συντονιστές. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε σήμερα μαζί μας.